Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα 7 λεπτά. Όμως είχα μια συνομιλία με μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου και γι' αυτό καθυστέρησα τις την κατανόηση και τη συγγνώμη σας, τη συγχώρεσή σα. Έχουμε την ημερήσια διάταξη λοιπόν και ρωτώ εάν έχετε κάποια πρόταση για τροποποίηση. Όχι. Στο σημείο 12 επισημένο προβλέπετε στα διάφορα, προβλέπετε μια ανταλλαγή απόψεων για, τις προτιμησιακές, ε, για το προτιμησιακό εμπόριο με την Ουκρανία. Άλλες παρατηρήσεις δεν υπάρχουν από ό,τι βλέπω και πάω στο σημείο 2, τα πρακτικά. Ω συνήθως, εάν δεν εκφραστούν αντιρρήσεις έως το τέλος της συνεδριάσεως, εγκρίνονται τα πρακτικά. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ενστάσεις ή αντιρρήσεις. Προχωρώ στο σημείο 3 οι συνήθεις ανακοινώσεις. Την Επιτροπή μας μπορεί να παρακολουθήσει κανείς από το διαδίκτυο. Γι' αυτό λάβετε το υπόψη και να συμπεριφέρεστε αναλόγως. Καταγράφεται σε ένα κατάλογο η αλληλογραφία εφόσον σας ενδιαφέρει μπορείτε να την πάρετε από τη γραμματεία έχουμε τις ακροάσεις μας α, ολοκληρώσει με την κυρία Μάλστρομ πρώτα, η οποία εξασφάλισε την υποστήριξη της πλειονοψηφίας εδώ στην Επιτροπή, από μια κάποια ε, επιπλέον επεξεργασία. Με τον κύριο Χάν, με την κυρία Μογκερίνη επίσης έγινε η ακρόαση και συμμετείχαμε και στην ακρόαση με τον κύριο Μοσκοβισή. Ευχαριστώ όλους τους αδέλφους που έλαβαν μέρος στις ε, εργασίες αυτές. Για την Επιτροπή Εμπορίου, είχαμε πολύ σαφή έκφραση των θέσεών μας. Για την Ουκρανία, όπως είπα στο σημείο 12 εντάσσεται η συζήτηση του θέματος αυτού στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για, την, ε, ε, για το θέμα που έχουμε ήδη συζητήσει, την αναβολή δηλαδή της θέσης εφαρμογή της συνθήκης σύνδεσης, συμφωνίας σύνδεσης. Υπό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ή υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ξεκίνησε μία, ε, έγινε μάλλον μία μια συνάντηση στην Γενέβη από τις 22 στις 26 Σεπτεμβρίου όπου εξασφαλίστηκε συμφωνία ως προς την ε, δυνατότητα καταγραφής σε καταλόγους των προϊόντων που εντάσσονται στο η συζήτηση. Προχωρούμε προς τον τρίτο γύρο για την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα ο ΠΟΕ έκανε ένα λεγόμενο public forum, μια δημόσια διαβούλευση την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε εκπροσώπηση από τέσσερις βουλευτές σε διάφορες ομάδες συζήτησης όπου ένα από μία από τις ομάδες συζήτηση αφορούσε συγκεκριμένα την συμμετοχή των ε, εκπροσώπων των κοινοβουλίων στην περίοδο μετά το Μπαλί και νομίζω ότι η δική μας παρουσία ήταν πολύ ισχυρή και ενίσχυσε, συνέβαλε στην ενίσχυση του διαλόγου του διακοινοβουλευτικού από τους εκπροσώπους των κοινοβουλίων των διαφόρων κρατών του κόσμου που συμμετέχουν στον ΠΟΕ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή στο πλαίσιο του φόρουμ του ΠΟΕ έγινε μια συνεδρίαση της Steering Committee, της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του ΠΟΕ, με εκπροσώπους της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Ενώσεως, IPU. Επικοδομητικό ήταν το ότι για άλλη μια φορά συζητήσαμε το θεματολόγιο για τη φάση μετά τον Παλή Είπαμε ότι δεν μπορούσαμε λόγω των αντιδράσεων ενός κράτους να εγκρίνουμε την, ε, τις προτάσεις για τον Trade Facilitator, οπότε πρέπει να ε, προχωρήσουμε στην επεξεργασία συγκεκριμένων θέσεων από τη Steering Committee, τις οποίες θα σας διανύμουμε. Έχουμε επίσης ακόμη, και θα το δείτε και στο πρόγραμμα, για τις 16 και 17 Φεβρουαρίου του 2015, την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΠΟΕ στην Γενέβη. Και τελευταία ανακοίνωση, θα το έχετε αντιληφθεί φαντάζομαι, ότι έχουμε τον ένατο γύρο για τις διαπραγματεύσεις για την ε, σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια ουσιώδη φάση, έχουμε ξεκινήσει μια ουσιώδη φάση των διαπραγματεύσεων. με στόχο να ολοκληρωθούν αυτές οι ε, διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες στις του 2015. Ο Πρωθυπουργό του Βιετνάμ θα είναι στις 13-14 Οκτωβρίου σε μια συνεδρίαση stock taking όπως ονομάζεται εδώ στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο Μπαρόζο για την καταγραφή των εξελίξεων και για τον προσδιορισμό των περαιτέρω βημάτων. Αυτά από μένα ως προς τις ανακοινώσεις και περνάω στο σημείο 4 που αφορά την κοινή συζήτηση για τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και κρατών μελών αφενός και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας αφετέρου μαζί με το θέμα της σύναψης συμφωνίας συνδέσης με την Μολδαβία. Αυτά αφορά η κοινή συζήτηση και δίνω το λόγο στον κύριο Μόησα, ε, εισηγητή μας. Παρακαλώ. Το μικρόφωνο δεν είναι αναμένο. Yes, we're okay now. Thank you, Chair. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έχουν καταθέσει τροπολογίες στην ομάδα της αυτή. Δύο κατηγορίες τροπολογιών υπάρχουν. Πρώτον, εκείνες που με κάνουν να ζηλεύω γιατί θα έπρεπε να τα είχα σκεφτεί εγώ αυτά που προτείνουν, η ομάδα μου τέλο πάντων, και εκείνες που μου φαίνονται ενδιαφέρουσες, αλλά πρέπει να τα συζητήσουμε πιο διεξοδικά σήμερα. Τι έχω ομαδοποιήσει τι τροπολογίε και θα ήθελα να σα παρουσιάσω τα κυρία σημεία του. Με... Παίρνοντα με τη σειρά τη πολιτικής ε, ομάδας και της σημασίας τους. Ο κύριος Κάσπαρη έχει προτείνει τρεις. Δύο από αυτές είναι από αυτές που με κάνουν να ζηλεύω. Είναι οι 15. Πράγματι δεν πρέπει απλώς να σημειώσουμε, πρέπει να ε, εκφράσουμε τη λύπη μας για τις ε, προβλήματα που δημιουργήσε στην ρωσική οικονομία οι, οι από τη Ρωσία. Η 15 πράγματι χρειάζεται η συμφωνία αυτή να εφαρμοστεί γρήγορα και αποτελεσματικά και επίσης θα πρέπει όπως λέτε στην τροπολογία 18 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ε, τη δυνατότητα να εξετάσει την εφαρμογή της. από τον κύριο Ζαχραντίν έχουμε λάβει διάφορες καλές τροπολογίες, οι πέντε που αναφέρει ότι μία από, ένα από τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει αυτή η Συμφωνία Σύνδεσης είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Τροπολογία 8 που αναφέρεται στο περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο θα βελτιωθεί με τη Συμφωνία Σύνδεσης, πράγματι. Πάντοτε όταν υπάρχουν προβλήματα στην οικονομία και ε, αβεβαιότητα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι πρώτες που πλήττονται, γιατί δεν έχουν τις, τους απαιτούμενους πόρους για να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα αυτή και το χάος που μπορεί να δημιουργηθεί. Υπάρχουν επίσης και κάποιες τεχνικές τροπολογίες που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάζει την εφαρμογή της συμφωνίας ε, είναι ξεκάθαρο ότι ο ρόλος του ότι αυτό θα γινόταν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά καλύτερα να είναι ακόμα πιο σαφές. Τροπολογία 16 από τον κύριο Ζαντό. Που αναφέρει ότι πράγματι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει τεχνική βοήθεια βράχει πρόθεσμα στη Μολδαβία έτσι ώστε να ε, καταφέρει να προσαρμόσει την ηθική της νομοθεσία και να υλοποιήσει τη συμφωνία. Ναι, είναι σωστό αυτό να το πούμε. Τώρα προχωρώ στις τροπολογίες του κυρίου Σούλτς. Εδώ είμαστε... Σόλτς, με συγχωρείτε. Ε, τροπολογία 2. Θα την υποστηρίξω. Πράγματι, χρειάζεται εμπειρογνώμονε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσουν τη δημόσια δίκηση τη Μολδαβία για την ε, υλοποίηση της Συμφωνία Σύνδεσης. Ωστόσο, οι άλλες τροπολογίε του κύριου Σόλτ δημιουργούν μια αντίποση που θα προσπαθήσω να σας περιγράψω με την οποία διαφωνώ και ελπίζω ότι και εσείς θα διαφωνήσετε. Σύμφωνα με τις τροπολογίες του κ. Σόλτς, λοιπόν, θα υποβάλουμε τη Μολδαβία σε θεραπεία σοκ. Ξαφνικά θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός με τρόπο ε, μη δίκαιο και θα ε, πλήξει αυτό κυρίως τις μικρομεσαίες ε, μολδαβικές επιχειρήσεις. Η υλοποίηση της Συμφωνίας Σύνδεσης θα υπονομεύσει τη δυνατότητα της Μολδαβίας να έχει δυνατή ισχυρή οικονομική θέση στην Ευρωασιατική ε, Ένωση, στην οποία υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή η Μολδαβία κατέχει σημαντική θέση και όλα αυτά θα έχουν δυσμενές επιπτώσεις στα δικαιώματα των Μολδαβών πολιτών. Θα σας αποδομήσω λοιπόν αυτές τις θέσεις του κ. Σόλτς. Τι μας λέει κατά βάση ο κ. Σόλτς ότι η Μολδαβία θα, πρέπει να, θα έπρεπε να συνεχίσει το οικονομικό μοντέλο που ακολουθεί το οποίο, κατά την άποψή του, είναι καλύτερο από εκείνο που της προτείνει της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με το επιχείρημα του, η Μολδαβία αποτελεί ένα αναπόσπαστο και, και καλά ενσωματωμένο στοιχείο του, της περιοχής εκείνων των κρατών που αποτελούσαν παλιά ε, τμήματα της Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτό όμως δημιουργεί ένα οικονομικό περιβάλλον χωρίς διαφάνεια, στο οποίο ε, ε, έχουν εξέχοντα ρόλο οι ολιγάρχες, δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία, η οποία διχάζεται, και αυτό οδηγεί και σε πολιτικές ε, πολιτικά προβλήματα όπως αυτά που έχουμε παρατηρήσει σε όλες περιοχές, σε άλλες χώρες της περιοχής μάλλον για να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση η Μολδαβία θα έπρεπε να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έρχομαι σε αυτό τον ισχυρισμό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει τη Μολδαβία σε σοκ. Θα γνωρίζετε ότι το 2001 έγινε μέλος του ΠΟΕ. Ο ΠΟΕ είχε επιβάλει χαμηλούς δασμούς όταν η Μολδαβία έγινε μέλος του. Το οποίο σημαίνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ένα τεράστιο, μια τεράστια αλλαγή προς την κατεύθυνση της φιλελευθερωποίησης της οικονομίας, γιατί ήδη η Μολδαβία είχε χαμηλού δασμού. Αναφέρεται επίσης και το θέμα της, της ασύμμετρης μεταχείρισης. Υπάρχουν κάποια προϊόντα που είναι ευαίσθητα για τη Μολδαβία, όπως τα γεωργικά και τα κλωστοϊφαντουργικά, για τα οποία θα ε, υπάρξει ειδική ρύθμιση. Αυτά έχουν ληφθεί υπόψη λοιπόν στη Συμφωνία Σύνδεση. Η μολδαβική οικονομία ήδη είναι ανοιχτή στον ανταγωνισμό. Αυτό που θα γίνει με τη Συμφωνία σύνδεση είναι ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη σύγκληση στον τομέα των υπηρεσιών και του κανονιστικού πλαισίου Πράγμα που θα δώσει τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στην ε, Μολδαβία. Δεν βλέπω λοιπόν πώς μπορεί να ε, βλάψει αυτή η συμφωνία ε, τους, τη μολδαβική οικονομία, τις μολδαβικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι είναι ήδη ανοιχτή η οικονομία, δεδομένου ότι προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος 8 ετών και οι μολδαβικέ επιχειρήσει, για παράδειγμα στον τομέα των γεωργικών και, ε, προϊόντων και των τροφίμων, στον οποίο έχει ένα ε, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η Μολδαβία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη ε, δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Γιατί αυτό να βλάψει τη Μολδαβία όσον αφορά τις επιπτώσεις στην κοινωνία από αυτή τη Συμφωνία Σύνδεσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια αξιολόγηση αντικτύπου, η οποία δείχνει ότι θα αυξηθεί το μέσο ε, ημερομίσθιο κατά περίπου 3% μέσω πρόθεσμα. Και προβλέπεται ότι οι μεταβολές στις, στην κατανομή των, ε, της δύναμης της εργατικής δεν θα ε, ξεπεράσει το 5% από τον ένα τομέα στον άλλο. Επίσης θα υπάρξει μια μικρή αύξηση των τιμών των γεωργικών προϊόντων, αλλά αυτό θα βοηθήσει και τους Μολδαβούς ε, γεωργούς, γιατί είναι ένας τομέας στον οποίο η Μολδαβία είναι ισχυρή και αν θυμάμαι καλά το 36% της, ε, του ΑΕΠ της Μολδαβίας είναι από τη γεωργία, είναι μια γεωργική οικονομία και εκεί προβλέπουμε μια αύξηση περίπου 5,4%. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι η Μολδαβία θα πρέπει να υιοθετήσει το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το δικό της ρυθμό. Εκείνη θα επιλέξει με ποια ταχύτητα θα το κάνει. Και αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξουν και ο τρόπος με τον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσει στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Θα έρθουν πιο κοντά στον ευρωπαϊκό ε, τρόπο ε, ε, λειτουργίας. Και δεν βλέπω κατά κανέναν τρόπο πώς αυτό θα μπορούσε να είναι κακό. Ίσως κάποιες επιχειρήσεις κάποια στιγμή χρονική να αντιμετωπίσουν το δίλημα αν προτιμούν να εστιάσουν περισσότερο στην ευρωπαϊκή αγορά ή στη μολδαβική αγορά, αλλά θα έχουν την ελευθερία να επιλέξουν ό,τι θέλουν. Ο κύριος Σόλτς επίσης ε, αναφέρεται στις σχέσεις της Μολδαβίας με άλλες ε, χώρες της Ευρωασιατικής Ένωσης και κατά βάση μιλάμε για τη Ρωσία. Ας μην ξεχνούμε όμως τι έγινε στην Ουκρανία και πώς η Ρωσία κινήθηκε στον οικονομικό τομέα έναντι της Ουκρανίας. Αυτές οι συμφωνίες σύνδεσης που δημιουργούν ζώνες ελευθερών συναλλαγών με τρίτες χώρες είναι συμφωνίες που γίνονται μετά από τη μερίδια πραγμάτευση, που γίνονται μετά από την ελεύθερη βούληση των κρατών να τις επιλέξουν που εκφράζεται ε, δημοκρατικά και από τις δύο πλευρές. Είναι λοιπόν λάθος να ισχυρίζεται κανείς ότι προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει στη Μολδαβία με γεωπολιτική επιλογή. Αντιθέτω, η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Μολδαβίας και οι δημοκρατικά εκλεγμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελευθερώ επιλέξει να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αποκόψει τη Μολδαβία από τρίτε αγορές. Είναι οι εμπορικοί εταίροι της Μολδαβία που θα το κάνουν. Πιθανώς. Επιβάλλοντας πιθανώς κυρώσει για να ε, τις δείξουν πόσο εξαρτημένοι είναι από εκείνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινείται έτσι. αντιθέτω, αυτό που έχουμε εδώ είναι μια ελεύθερη επιλογή. Σα ευχαριστώ και ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις ε, συναδέλφων αν θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, με άλλα λόγια αντιτίθεμε σε όλες τις τροπολογίες του κυρίου Σόλτς με την εξαίρεση της τροπολογίας 2 αν θυμάμαι καλά. Ναι, η 2. Αυτή μπορώ να την ε, αποδεχτώ και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα για τους σκιώδεις. Ο κύριος Βίνκλερ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την εισηγησή του και για το έργο το οποίο επιτέλεσε για το θέμα αυτό. Και θα έχουμε κάποιες τροπολογίες. Και θα πρέπει να ξεχνούμε σε σχέση με την δραστηριότητα των τελευταίων ετών ότι εδώ στην Επιτροπή μας το τελευταίο τριετη τριετή-τετραετή έχει ξαναζητηθεί το τι θα γίνει με την ε, Μολδαβία. Βέβαια τα πράγματα γίνουν πιο ευχάριστα, πιο ευχάριστα από ό,τι ισχύει στην ε, Γεωργία, στην Ουκρανία, σε άλλους εταίρους μας της Ανατολικής Ευρώπης. Οπότε η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το, τελευταίο μήνα έχουν εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας εκείνους και έτσι προσπαθούμε κάτι να κάνουμε όσον αφορά με τα όσα συμβαίνουν στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το Κοινοβούλιο στην μεγάλη του πλειοψηφία προχωρεί προς ε, μια ταχεία σύνοψη αυτής της συμφωνίας Και αυτό θα αποτελεί ένα μήνυμα. Ότι τα κρατη θα πρέπει να κυρώσουν αυτή τη συμφωνία. Βέβαια, για τις αποφάσεις μας έχει μετρήσει η πολιτική συγκυρία. Έχουμε τώρα και το θέμα των εκλογών στη Μολδαβία της 30 Νοεμβρίου. Είναι λιγότερο από δύο μήνες. Οπότε, οι πολιτικές ομάδες συμφωνήσουν και εδώ, αν επιψηφίσουμε το κείμενο, ελπίζω να εγκριθεί η γνωμοδότηση αυτή και στην Ολομέλεια. Οπότε έτσι θα μπορέσουμε να στείλουμε αυτό το αποφασιστικό πολιτικό μήνυμα και στη Μολδαβία και στους άλλους εταίρους μας. Χαίρομαι που η αναπτυξιακή συμφωνία έχει ταχαίως τεθεί σε λειτουργία. Ακριβώς γι' αυτό και λέω ότι τελευταία διετία, τριετία τουλάχιστον εδώ στην Επιτροπή μας συμφωνούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και να συνάψουμε αυτή τη συμφωνία με την Μολδαβία κατά το Ευρωπαϊκό Τμήμα. Τώρα για τις τροπολογίες τις έχω μελετήσει να μην ασχοληθώ μία-μία με τις τροπολογίες αλλά το ΕΛΚ συμφωνεί με εκείνες οι οποίες συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή προσέγγιση ούτως υπήν για την Μολδαβία. Ο πρόεδρος και κυρία Αντιπρόεδρε σας ευχαριστώ. Τώρα ο άλλο αντιπρόεδρος μας, ο κύριο Ζαχράντιλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Επικέντρο του ενδιαφέροντό μας η Δημοκρατία τη Μολδαβία εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε γι' αυτό και θέλουμε να την εντάξουμε στο θεσμικό μας πλαίσιο. Οπότε γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό έχουμε αυτή η έκθεση. Οπότε δεν μπορούμε παρά να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για τον υπεύθυνο και ολοκληρωμένο τρόπο με τον οποίο δούλεψε. Ελπίζω θα ψηφίσουμε ακριβώς όπως εκείνος μας συνέστησε. Θα έπρεπε να είναι όλοι ρένα, αλλά εν πάση περιπτώσει, Ναι, όντως ομιλώ εκ μέρους του όλοι ρένα, αλλά και γενικότερα εκ μέρους της ομάδας Άλντε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή και τους συναδέλφους για την επικοδομητική συνεργασία. Οι διαπραγματεύσεις με τη Μολδοβία ήταν αρκετά δύσκολες γιατί διανύσαμε τρεις διαφορετικές κυβερνητικές κρίσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ίσως χρειαστεί και το Νοέμβριο να αντιμετωπίσουμε νέες και περίπλοκες συνθήκες μετά τις νέες εκλογές. Ε, πάντως ε, υπάρχουν σημαντικά βήματα για νέες οικονομικές εξελίξεις και σε δύσκολες οικονομικά περιόδους. Μπορούμε με την ε, ε, συνεργασία αυτή να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής για τους πολίτες. Εν γέννη το εμπόριο έχει συμβάλει σε περισσότερη ευημερία σε πολλές χώρες και θα πρέπει να διατηρήσουμε την αισιοδοξία μας ότι η τάση αυτή θα ισχύσει και για το μέλλον και θα προσφέρει νέα ευημερία για τους πολίτες της Μολδαβίας που είναι μια ακόμα από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης. Επίσης, με τη συμφωνία αυτή μπορούμε να έχουμε νέες δυνατότητες επέκτασης και συνεργασίες σε νέες αγορές. Καταργούνται αυτομάτως δασμοί σε πολλά προϊόντα και Διατηρούνται βέβαια κάποια προβλήματα, παραμένουν κάποιες προκλήσεις που σημαίνουν καταρχάς την υλοποίηση της συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή μπορεί να έχει νόημα μόνο εάν εφαρμοστεί σωστά από τις δύο πλευρές, όπως άλλωστε κάθε συμφωνία. Μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση των, ε, του, της πολιτικής, της εμπορικής και των πολιτικών και των διατάξεων της Μολδαβής προς το εμπόριο με βάση και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σημαίνει τη δυνατότητα για μέσα εξωτερικές επενδύσεις στη χώρα και μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο προβλέψιμο θετικό περιβάλλον για τους επενδυτές και τις εμπορικές σχέσεις. Οι συνομιλίες με τη Μολδαβία θα πρέπει να προωθηθούν με στόχο την απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών, ακόμα μερικά καλά παραδείγματα ε, όπου ο ελεύθερος ανταγωνισμός φέρνει καλά αποτελέσματα. Τα έχουμε δει στο χώρο της ενέργειας. Η Μολδαβία, η οποία εξαρτάται 100% από το μονοπόλιο του φυσικού αερίου της Γκάσπρο έχει προχωρήσει στην πρώτη φάση της σύνδεσης με τον ε, με το μηχανισμό σύνδεσης ε, του αγωγού από τη, Ρωμανία, από τη Ρουμανία και έτσι μπορεί να έχει την ελπίδα για πιο φθηνό ε, φυσικό αέριο. Γιατί τώρα πληρώνει την πιο ακριβή τιμή στο φυσικό ε, αέριο με 380 δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Helmut Σόλτ, Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την ανοιχτή του τοποθέτηση ως προς τις δικές μας ε, τροπολογίες. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω τα εξή προκαταβολικά, ότι ναι, έχουμε αντίληψη του γεγονότος ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κεφάλαιο, μια συμφωνία συνδέσεως, η οποία θα έχει σημαντικές συνέπειες για τη μολδαβική οικονομία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Ακριβώς εδώ είναι η πτυχή την οποία προσπαθούμε να επισημάνουμε στο σχέδιο της εκθέσεως, της γνωμοδότησης του συντάκτη για να επισημάνουμε τις συγκεκριμένες συνέπειες βράχη και μέσο πρόθεσμες προοπτικές για τους πολίτες της Μολδαβίας δεν έχουμε καταστήσει σαφέ ότι δεν έχουμε δηλώσει δηλαδή ότι εν γέννη το εμπόριο με τη Μολδαβία είναι απορριπταίο ή ότι δεν θέλουμε την σύνδεση. Διότι εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφής δήλωση βούλησης της πλειονότητας του μολδαβικού λαού. Η Μαρίτσια το επεσήμανε. Έχουμε ε, διανύσει μια περίοδο με τρεις κυβερνητικές αλλαγές. Μια περίοδο κυβερνητικών κρίσεων ε, αλλεπάλληλων και εδώ η θέση της Μολδαβίας και στο παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό είναι ζήτημα δημόσιου διαλόγου. Πρέπει λοιπόν με πολύ μεγάλο αίσθημα υπευθυνότητας να ελέγξουμε και να επαληθεύσουμε τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η συμφωνία για τους πολίτες ακριβώς επειδή επίκυνται και εκλογές τώρα τον Νοέμβριο. Και αυτό σημαίνει ότι βεβαίως δεν θέλουμε να λησμονηθεί το θέμα αυτό από το δημόσιο διάλογο στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι είναι σε σχέση με την τροπολογία 14 διότι εδώ εμεί καθιστούμε απόλυτο σαφέ ότι ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ανησυχούμε για τις βράχοι και μέσο πρόθεσμες συνέπειες της εφαρμογής της συμφωνίας για την κοινωνική και οικονομική ζωή των πολιτών της Μολδαβίας και ιδιαίτερα όσον αφορά την απασχόληση. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι σε χώρες όπως η Μολδαβία που έχουν μέσο εισόδημα 100 ευρώ θα υποστούν τέτοιου είδους χώρες τεράστιες συνέπειες από την εισαγωγή αυτής της ε, συμφωνίας λόγω της ε, ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης των ευρωπαϊκών προϊόντων στην εσωτερική του αγορά. Και άρα πιστεύω θα πρέπει με μεγάλη υπευθυνότητα να χειριστούμε τα θέματα αυτά για το θέμα της υπερθυμιστερίας. Με προβληματίζουν αυτά τα οποία λέει ο εισηγητής, ο συντάκτης και γι' αυτό θα ήθελα ε, να αξιολογήσει πιο προσεκτικά τις τροπολογίες μου τις σχετικές. Εμείς ως ομάδα εν γέννη εξετάζουμε μεγάλη προσοχή της ε, τροπολογίας των λοιπόν συναδέλφων και ομάδων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, βλέπω ότι δεν υπάρχει από τους πράσινους και όδης. Α, ο Γιάννικ είναι εδώ. Συγχαρητήρια, είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η δουλειά του εισηγητή και θα θέλαμε πάρα πολύ κάποιοι από τους υποψήφιους ε, επιτρόπους να έρχονται και εκείνοι το ίδιο σοβαρά προετοιμασμένοι εδώ στις Επιτροπές για τις Ακροασίες όσον αφορά το κείμενο καθε αυτό για τους οικολόγους, για τους πράσινους. Αυτές οι συμφωνίες είναι κάτι το μπερδεμένο γιατί βεβαίω και είμαστε επί της αρχής υπέρ αυτών των συμφωνίων σύνθεσης, αλλά έχουμε αυτή την προσέγγιση στο κοινωτικό κεκτημένο το οποίο ε, ακολουθεί. Όμως θέλουμε να υπάρχει δημοκρατία, κράτος δικαίου, όπως πάντοτε προϋποτίθεται για αυτές τις συμφωνίες, αλλά, αλλά από την άλλη μεριά εμείς θεωρούμε ότι το κίνητρο είναι εμπορικό εμπορικό κέρδο και γι' αυτό και η επιθυμία πάντοτε είναι να προχωρήσουν γρήγορα αυτέ τις συμφωνίε και βεβαίω θα έχουμε κάποιες τροπολογίε. όσον αφορά το κόστος της προσαρμογής, το βραχυπρόθεσμο που θα πρέπει να φέρει η οικονομία της χώρας, να δούμε επίσης και τις κοινωνικές επιπτώσεις. Μια που Έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση υπάρχει ένα κοινωνικό κόστος στην προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, la ringrazio per il suo lavoro. Ε, noi siamo fondamentalmente. Σας ευχαριστώ. Βασικά, εμείς συμφωνούμε με όλα όσα είπατε. Πάντω θα ε, υπάρξουν θετικές επιπτώσεις ε, για την ε, μολδαβική κοινωνία, κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Βεβαίω και η Ένωση ζητεί μεταρρυθμίσει από τι χώρες που βρίσκονται εκτό. Ένωσης, αλλά είναι όμορε. Και θα πρέπει να δούμε τι προβλήματα τυχόν θα προκύψουν. Κύριε Σόλτ, πολύ σύντομα παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μια ακόμα πτυχή που λησμόνησα νωρίτερα είναι σημαντική, μια και την έθιξε και ο συντάκτη. Έχουμε εδώ να κάνουμε με τι οικονομικέ σχέσει στην Ευρασιατική Ένωση. Ε, εδώ πέρα στι τροπολογίε που έχω καταθέσει, ιδιαιτέρω με ενδιαφέρει να αναζητηθεί ένα τρόπο με τον οποίο η παραδοσιακή οι παραδοσιακοί οικονομικοί δεσμοί που έχει η Μολδαβία με τις ε, χώρες αυτές ε, και με τις οποίες έχουμε και συμφωνίες σύνδεση όπως η Ουκρανία και η Μολδαβία θα διαφυλαχθούν, δεν θα ανατραπεί δηλαδή η οικονομική σχέση με την Ευρασιατική Ένωση, περιλαμβανομένης βέβαια και της ε, ε, Ρωσικής ε, Άρα θα πρέπει να μην είναι εμπόδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοιου είδους σχέσεις. Δεν θέλουμε μόνο μονομερή σχέση με προϋποθέσεις, είτε αυτό είτε τίποτα, αλλά έναν διάλογο για τις οικονομικές σχέσεις και με την Ευρασιατική Ένωση αυτών των κρατών. Είναι ένα σημείο το οποίο νομίζω θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ προσεκτικά. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν, θα έκανε άλλο το λόγο, οπότε θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το εμπορικό σκέλος της Συμφωνίας Σύνδεσης την οποία σας υποβάλλουμε, η DCFTA, πιστεύω ότι ο εισηγητής έχει συνοψίσει επαρκώς την κατάσταση. Όσον αφορά τις ανησυχίες τώρα που έχουν εκφραστεί οι το ότι η Μολδαβία θα υποβληθεί σε μια θεραπεία σοκ. Η Μολδαβία θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα ε, ορισμένους τομείς, τους οποίους θα προστατεύσει ιδιαίτερα, ε, πιο συγκεκριμένα τα γεωρικά προϊόντα Θα μπορούσαμε να πούμε ότι για πρώτη φορά η Μολδαβία θα έχει σε τέτοιο επίπεδο δυνατότητα πρόσβαση στην υπηγορά υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, δεν δέχομαι ότι θα υπάρξει σοκ. Ίσως υπάρξουν προσαρμογέ, αλλά σε καμία περίπτωση σοκ. Θα υπάρξει επίση και τεχνική βοήθεια προ τη Δημοκρατία τη Μολδαβία στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Έχει προβλεφθεί ε, στη διάρκεια τριών ετών περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ ένας προϋπολογισμός προς αυτήν την κατεύθυνση και για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για την υποστήριξη λοιπόν και την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι με αυτή τη συμφωνία θα ε, εξυγχρονιστεί η οικονομία της ε, Μολδαβίας και θα δημιουργηθεί μια εις βάθος ζώνη ελευθέρων συναλλαγών Αναφερθήκατε επίσης και σε πολιτικές ε, λιτότητας. Εγώ θα έλεγα ότι εδώ εστιάζουμε σε εμπορική πολιτική της Μολδαβίας. Τώρα όσον αφορά τις σχέσεις με την Ευρωασιατική Ένωση και τη Ρωσία, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στην συνθήκη η οποία να απαγορεύει στην Μολδαβία να συνεχίσει να έχει μια προνομιούχα σχέση με τη Ρωσία ή με άλλους εμπορικούς εταίρους, κάθε άλλο. Αντιθέτως όμως διαπιστώνουμε ότι η Ρωσία είναι εκείνη που επέλεξε να επιβάλλει εμπορικούς ε, φραγμούς, εμπάργκο στα μολδαβικά γεωργικά προϊόντα. Επομένως δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που προκαλεί αυτές τις ε, κυρώσεις, είναι ε, επιλογή της Ρωσίας για να ασκήσει πίεση στη Μολδαβία. Τώρα όσον αφορά την υπερτινιστερία. Εδώ και τρία χρόνια έχουν ξεκινήσει ε, συζητήσεις ε, με τους εκπροσώπους της υπερνηστερίας. Έχουμε επευθυνθεί προς αυτούς. Ανταποκρίνονται και θα συνεχιστούν αυτές οι ε, συζητήσεις. Από το 2015 που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται αυτές οι, αυτά τα μέτρα προνομιακής ε, μεταχείρισης θα μπορεί να επωφεληθεί και η υπερδνηστερία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν προσπαθεί να επιβάλλει τις θέσεις της, αντιθέτως προσπαθεί να έχει μια σχέση ε, συζήτησης και διαλόγου ε, με την ε, πρόσωπο της περιοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και συντομότατα ο εισηγητής. Λοιπόν, σε δύο σημεία εγώ θέλω να αναφερθώ. Η υπερδνηστερία πρώτον και δεύτερον η Ευρωασιατική Ένωση και γέφυρες με αυτήν. Πρώτον, όσον αφορά την υπερδνηστερία, αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει την εθνική κυριαρχία της Μολδαβίας στην περιοχή αυτή. Γιατί οι οικονομικοί φορές, φορείς, οι πολιτικοί φορείς, οι επιχειρήσεις της υπερδνηστερίας θα επιθυμούν να εποφεληθούν από αυτή τη συμφωνία σύνδεσης και αυτό θα τους αναγκάσει να αποδεχθούν τους μολδαβικούς κανόνες. Άρα θα έλεγα ότι αντιθέτως δεν ε, περιπλέκει τα πράγματα, ενισχύει τη θέση του Κισνάου ε, και την ε, ε, κυριαρχία του υπερθυνιστερίας επίσης. Όσον αφορά τώρα το, τη δημιουργία ε, σχέσεων και την Ευρωσυντική Ένωση. Δεν είμαστε εμεί αυτοί που γκρεμίζουμε τι γέφυρε. Αντιθέτω, εμεί του διευκολύνουμε να χτίσουν γέφυρε. Τώρα, εάν η Ρωσία επιλέγει ε, να επιβάλλει κυρώσει για να ασκήσει πίεση στη Μολδαβία, δεν πρέπει εμεί να θεωρούμε ότι η ευθύνη βαρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάποιε κάποιες βασικές αρχές στον δυτικό πολιτισμό, την, ελεύθερη, την ελευθερία, ε, τη δυνατότητα να επιλέγουμε ελεύθερα τι πράττουμε Εάν κάποιο προσπαθεί να ασκήσει πίεση για να μην ε, επιλέξουμε ελεύθερα αυτό που επιθυμούμε, δεν φταίμε εμεί. Η Μολδαβία, αν θέλει να συνεχίσει να έχει προνομιακέ σχέσει με του παραδοσιακού τη εταίρου, μπορεί να το κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να έχει ε, καλέ εμπορικέ σχέσει με τη Ρωσία, με την προπόθεση βέβαια ότι η Ρωσία ε, σέβεται το διεθνέ δίκαιο και του κανόνε του ΠΟΕ. Πώ θα μπορούσαμε εμείς, όταν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε την επιθυμία να σταματήσουμε τις σχέσεις μας με τη, τις εμπορικές με τη Ρωσία, πώς θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από μια τρίτη χώρα, εν προκειμένου τη Μολδαβία, να σταματήσει να περιορίσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Επομένως όλο αυτό το, το επιχείρημα δεν στέκει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα λοιπόν. Πρώτη συζήτηση 24 Σεπτεμβρίου, τροπολογίες έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γίνεται η ψηφοφορία και στις 16 Οκτωβρίου ψηφίζει η Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων για να πάει το θέμα αυτό στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο, όπου θα γίνει η οριστική ψηφοφορία, η τελική ψηφοφορία. Και τώρα περνάω στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το υπαριθμό 6. που έχει να κάνει με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο. Ο Γκραφ Λάμπστορφ δεν είναι εδώ. Ο Μαρίτσια, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό ο μέρους του Αλεξάνδρου Λάμπστορφ. Ε, σε αυτό το σημείωμα και έχει το σχέδιο της ε, έκθεσης του τεχνικού χαρακτήρα όσον αφορά τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφει το 1992 ε, και κυρώθηκε το 1994 αλλά σύμφωνα με τις σημερινές εκτιμήσεις η Κροατία αναλαμβάνει να προσχωρήσει σε αυτήν την ε, συμφωνία που αφορά τον ΕΟΧ και ε, όσον αφορά τη συμμετοχή της χώρας έχουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου ούτω ώστε να αυτή τη συμφωνία για την συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον ΕΟΧ και έτσι θα υπάρχει θα, προ, προσφοράψει και το πρωτόκολλο για, με, την Νορβηγία για την περίοδο 2009-2014 κατόπιν της συμμετοχής της ε, Δημοκρατίας της Κροατίας στον ΕΟΧ. Θα έχουμε το επιπλέον πρωτόκολλο ε, το οποίο θα, αυτό το πρόσθετο πρωτόκολλο μεταξύ Ισλανδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο προσχωρεί η Κροατία και τέτοιο υπάρχει το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας ε, με την Νορβηγία που και εκεί θα προσχωρήσει η Κροατία μετά την προσχώρηση στον ΕΟΧ. Εδώ έχουμε τα τρία μέλη της ε, ΖΕΣ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, ε, Νορβηγία και, στο, και, και τις χώρες του ΕΟΧ, όλα δηλαδή τα κράτη-μέλη, σε μια ενιαία αγορά και εδώ έχουμε μια ε, νομοθεσία και έχουμε τις τέσσερις ελευθερίες για πρόσωπα, ε, κεφάλαια υπηρεσία σε αγαθά, την ελεύθερη κυκλοφορία του επίση καλύπτεται εδώ πέρα και η παιδεία, κοινωνική πολιτική, έρευνα, περιβάλλον, ε, καταναλωτέ, τουρισμό, πολιτισμό, όλα αυτά που ονομάζουμε συνοδευτικέ οριζόντιε πολιτικές και η συμφωνία εξασφαλίζει ίσα δικαιώματα υποχρέωση στην εσωτερική αγορά για του πολίτε και του οικονομικού φορεί. Ο εισηγητή πρεσβεύει το ότι η συμμετοχή τη Κροατία στον ΕΟΧ είναι συνέπεια φυσική της προχώρησή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι αυτονόητο το ότι πάνω από ένα χρόνο δεν προσχώρησε. Ε, Επιτροπή και Συμβούλιο έχουν λάβει τα μέτρα ούτω ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμμετοχή στον ΕΟΧ. Ε, βάσει όλων αυτών ο ε, προτείνει να εγκρίνεται αυτό το τεχνικό κείμενο. Ευχαριστώ λέει και τώρα ο λόγος στους σκιώδεις εισηγητές. Not... Ah, Είστε εδώ, όχι, ο Ντέβιτ Μάρτιν. Κώστας Μαυρίτης είναι ο δικός μας ο δεν μπόρεσε να παραστεί και μου έστελε ε, ένα κείμενο και εν συντομία λέει ότι είναι τεχνικό χαρακτήρα το κείμενο και δεν έχουμε ε, κάποια ένσταση και οι σοσιαλιστές πρόκειται να εγκρίνουν το κείμενο. Ε, ECR, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Ζαχράντελ, όπως πάντα. Σχεδόν είμαι θα υποχρεωμένη να ολοκληρώσουμε την ε, ευρωπαϊκή πορεία της Κροατίας. Οπότε δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με την πρόταση του εισηγητή για την συμμετοχή της χώρας στον ΕΟΧ και στις τρεις συναφείς συμφωνίες. Ο κύριος Κατρούγκαλος για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά. Ο κύριος Κατρούγκαλος έχει το λόγο. Support, uh, the proposal. Συμφωνούμε με την πρόταση. Mr. Borelli, EFD. EFD. Oh. Εκτός μικροφώνου. Δεν ακούστηκε τι είπε ο βουλευτής της ε, EFD. Τώρα ο πρόεδρος είναι εκτός μικροφώνου. Α, Α, συμπαθάτε με λέει. Έχει ζητήσει άλλο το λόγο. Όχι, επομένως τώρα να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Νίτα. Good morning everyone. Uh, I'm here. the Κυ κύριος. Σας ευχαριστούμε για την σύμφωνη γνώμη σας όσον αφορά την ε, εκθεσή μας παρέλθε ένα χρόνο από την προσχώρηση τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εσήμανε η ώρα, ούτω ώστε και η χώρα ε, αυτή να γίνει ε, πλήρε μέλο ει ε, την συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Θα ο εισηγητή ή η εισηγήτρια. σα σας ευχαριστούμε, καλύφθηκα, λέει η εκπρόσωπος του εισηγητή. Θα ψηφίσουμε στις 10 Οκτωβρίου μέχρι τις 5 Νοεμβρίου οι τροπολογίες και στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου πρόκειται να γίνει η τελική ψηφοφορία. Τώρα έχουμε τις ψηφοφορίες. Α, όχι, όχι. Έχουμε την παρακολούθηση των ομάδων. Στους συντονιστές συζητήσαμε αυτές τις ομάδες που αποτελούν μια καλή πρακτική των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες του κόσμου και είπαμε ότι θα είναι καλό να συνεχιστεί αυτή η πρακτική αλλά και να θεσπιστούν νέες εγκάρσιου χαρακτήρα, ε, ε, τον οποίο βέβαια θα πρέπει να προσδιορίσουμε και τα χαρακτηριστικά. Τώρα, έχουμε σχεδόν όλους τους μόνιμους εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές από τις πολιτικές ομάδες θα κοινοποιηθούν σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, μάλλον κοινοποιήθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου τα ονόματα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, προκειμένου να ε, επικρατήσει διαφάνεια. Μόνο η ομάδα παρακολούθησης σε σχέση με τις ΗΠΑ έχει συνεδριάσει μέχρι τώρα, όμως προβλέπονται ακόμα δύο στο χρονοδιάγραμμά μας. Μία που προβλέπεται για σήμερα συγκεκριμένα για το Βιετνάμ και μία για αύριο που θα ασχοληθεί με το Εκουαδόρ και την προσχώρηση στη Συμφωνία Κολομβίας-Περού. Η ομάδα παρακολούθησης για τις Ηνωμένε Πολιτείες συνεκλήθη τάχιστα προφανώς λόγω των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία TTIP της προηγούμενης εβδομάδας και έτσι στις 25 Σεπτεμβρίου έγινε μια προκαταρκτική ενημέρωση στην ομάδα αυτή παρακολούθησης Monitoring Group για τις εξελίξεις που διαγράφονταν στον έκτο γύρο διαπραγματεύσεων της Washington κατέστη σαφές εκεί ότι ορισμένα κεντρικού χαρακτήρα ζητήματα περιεχομένου που θα έπρεπε να συζητηθούν δεν περιλαμβάνονται. Φερρυπίν το ζήτημα των δημοσίων προμηθειών. ζητήθηκαν όμως άλλα ζητήματα ρυθμιστικού χαρακτήρα και μπορούμε να πούμε μετά το νέο γύρο διαπραγματεύσεων της Ουάσιγκτον ότι η συζήτηση που είχε γίνει στην ομάδα παρακολούθησης ήταν εύστοχη, είχε τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς να είναι ούτε αποτυχημένη ούτε ρηξικέλευθη, απετέλεσε μια συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Η πλήρης ενημέρωση για το γύρο των διαπραγματεύσεων θα γίνει στην ομάδα παρακολούθηση την προσεχή εβδομάδα, ώστε και αυτή η ομάδα παρακολούθηση της σχέσης των ΗΠΑ ε, να είναι ενήμερη. Οι άλλες επίσης ομάδες παρακολούθησης συγκαλούνται ως ήθιστε όταν προκύπτουν ζητήματα στο πρόγραμμα, στο χρονοδιάγραμμα που τις αφορούν. Στον επόμενο γύρο πιστεύω θα πρέπει να δούμε εάν είναι όντως εύστοχη η λειτουργία και οι επιλογές ε, εργασίας των ομάδων αυτών σε σχέση με τις διαπραγματεύσει. Αυτά έχω να πω εγώ από πλευράς μου και ρωτώ, Χέλμουτ, εάν έχετε κάτι να πείτε κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, ο κύριος Σόλτς. Ε, θα ήθελα απλώ να ενημερώσω ότι αύριο στι 10 έχουμε την ομάδα παρακολούθηση για το Εκουαδόρ. σα το λέγω γιατί θέλω να είναι παρόντε όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι τη Επιτροπή μα σε αυτή την ε, πολύ σημαντική συνεδρίαση τη ομάδα παρακολούθηση. Και επίση θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχετε πιο συγκεκριμένε πληροφορίε για την ε, διεξοδική ενημέρωση για την έκβαση αυτού του έκτου γύρου διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον για την Επιτροπή παρακολούθηση με τι ΗΠΑ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είναι το εξή. Είτε την Τρίτη είτε την Τετάρτη τη προσεχικού εβδομάδα θα έχουμε το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα. Μέχρι στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Κύριε Ζαχράντιλ. Χαίρομαι για το γεγονό ότι θα γίνει αυτή η πρώτη συνάντηση τη ομάδα παρακολούθηση μετά τι εκλογέ ε, τι ευρωπαϊκέ, αμέσω μετά τη συνάντηση τη Επιτροπή μα σήμερα. Ευχαριστώ. Καλώς, δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Δέκα είναι η ώρα. Εν τη αυτή ξεκινάει ο γύρος των ψηφοφοριών και σας υπενθυμίζω ότι χρειάζεστε όλη την κάρτα σας, την ηλεκτρονική για την ψηφοφορία. Οι πολιτικές ομάδες φαντάζομαι θα περιοριστούν στον αριθμό των ψήφων που διαθέτουν στην Επιτροπή. Και προχωρώ στο πρώτο θέμα για ψηφοφορία που είναι η Συμφωνία Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. ψηφοφορία ηλεκτρονική και μοναδική. Άρχεται. Πέρας. 36 ψήφισαν. 29 υπέρ, μία αποχή, 5 ψηφικάτα Η επόμενη ψηφοφορία πάλι αφορά την ε, σύναψη της συμφωνίας ε, σύνδεσης με τις λοιπές με τα λοιπά τμήματα, όχι δηλαδή την ε, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και ψηφίζουμε την τροπολογία 13 παραγράφους 1 του κύριου Σόλτς σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Όχι ηλεκτρονικά. Διανατάσεως της χειρός. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Παράγραφος Τροπολογία 14 για την παράγραφο 2. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 15 του κύριου Κάσπαρη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 του κυρίου Ζαντό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 του κυρίου Κάσπαρη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 του κυρίου Κασπάρη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 Ζαχράντι Λιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 παράγραφος 4α νέα του κύριου Σόλτς υπέρ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία πρώτη για την αιτιολογική σκέψη α υπέρ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 2 για νέα αιτιολογική σκέψη ΑΑ του κ. Σόλτς υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Τροπολογία 2 του κ. Σόλτς. Πέρας της ψηφοφορίας. υπέρ 16 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 3 του κυρίου Σόλτς υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 4 του κυρίου Σόλτς υπέρ. κατά αποχές απερίφθη Πέντε του κυρίου Ζαχράντη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 του κυρίου Σόλτς υπέρ κατά αποχές απερίφθη Τροπολογία 7 του κυρίου Σόλτς υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 8 του κυρίου Ζαχράντη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 του κυρίου Σόλτς. Υπέρ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 10 του κύριου Σόλτς υπέρ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 11 του κυρίου Μόησα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 12 του κυρίου Σόλτς υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά και ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. 32 υπέρ, μία αποχή, πέντε ψήφοι κατά. Και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έτσι ολοκληρώθηκε ο γύρος των ε, ψηφοφοριών για σήμερα και περνώ στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης νέα τρόφιμα. Δεν είναι από τα θέματα που πραγματευόμαστε καθημερινά στην Επιτροπή μας. Έχουμε να κάνουμε ένα καινοφανές θέμα στις ε, εμπορικέ διαπραγματεύσεις. Πάντως πρόκειται για ένα ζήτημα σημαντικό, για ένα σημαντικό ζήτημα, τα νέα τρόφιμα που θα διαδραματίσει και όλο, όλο και πιο έντονο ρόλο στις εμπορικές διαπραγματεύσει, Χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα τώρα να δώσουμε στην κυρία Ντάρλινγκ τον λόγο, την συγκεκριά μας. Uh, um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η γνωμοδότηση που συζητούμε σήμερα έχει σχέση με τον προτινόμενο κανονισμό για τα νέα τρόφιμα. Η αρμόδια επιτροπή είναι η ΕΝΒΗ περιβάλλοντος. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία για το ιστορικό, προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε το, το ρυθμιστικό πλαίσιο του κανονισμού που ισχύει αυτή τη στιγμή από το 1997. Έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο δίνεται η άδεια για την τοποθέτηση στην αγορά νέων τροφίμων. Ο στόχος είναι αυτή η διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσματική ε, διαφυλάσσοντας την ασφάλεια των τροφίμων. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να είσαστε ήσυχοι. Παρακαλώ, ησυχία. Okay. Um, ε, ωραία, ευχαριστώ λοιπόν. Όπω έλεγα, ο στόχο είναι η διαδικασία αυτή να γίνει πιο αποτελεσματική, διασφαλίζοντα ταυτόχρονα όμω, ότι τα πρότυπα ασφάλεια ε, τροφίμων θα είναι τόσο υψηλά όσο απαιτούν οι καταναλωτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα τρόφιμα είναι τρόφιμα τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν η ανθρώπινη κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τις 15 Μαΐου του 1997. Αυτό καλύπτει πολλά τρόφιμα τα οποία ε, περιέχουν για παράδειγμα ε, συμπληρώματα διατροφής, ε, νανοηλικά. Έμαθα ένα σωρό πράγματα για τα νέα τρόφιμα σε αυτή την γνωμοδότηση. Με την νέα της πρόταση όμως η Επιτροπή εξαιρεί τα κλωνοποιημένα τρόφιμα ή τα τρόφιμα τα οποία έχουν ε, δημιουργηθεί με επεξεργασία κλωνοποιημένων. Υλικών. Είναι η δεύτερη προσπάθεια για να αλλάξει το ε, ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτά τα τρόφιμα. Όσον αφορά τώρα την κλωνοποίηση, η η συγγήτρια έχει αντιληφθεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παρουσιαστεί μια νέα πρόταση ξεχωριστή της Επιτροπής ε, και ε, θα τη συζητήσουμε στην Επιτροπή μας και τότε με χαρά θα σας παρουσιάσω τη σχετική γνωμοδότησή μου. Θα προτείνουμε λοιπόν στην αρμόδια Επιτροπή να αποδεχθεί την πρόταση της, Επιτροπή, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμείς εστιάζουμε στα στοιχεία που ε, σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο. Υπάρχουν τα τρόφιμα εκείνα τα οποία είναι παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη χώρα, είναι τρόφιμα τα οποία ήταν συνήθι για τις τρίτες χώρες, απλώς είναι νέα για εμάς, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα τρόφιμα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να υπάρχουν επαρκείς ε, δικλείδας ασφαλείας. Εμείς υποστηρίζουμε, η εισηγήσή μου είναι να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθεια να δημιουργήσει μια διαδικασία ε, γρήγορη, fast track για τα τρόφιμα αυτά. Ωστόσο, όταν πρόκειται στην ευρωπαϊκή αγορά να δημιουργηθούν, να, να εμπορευτούν παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη χώρα, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν εμπόδια. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ξεκάθαρο ποιε πληροφορίε αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει από του παραγωγού αυτών των παραδοσιακών νέων τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή αναφέρεται σε ένα ιστορικό ασφαλούς χρήσης το οποίο να δείχνει ότι τα τελευταία 25 χρόνια ε, το τρόφιμο αυτό καταναλώνεται χωρίς προβλήματα. Η αρχές αυτές όμως είναι ε, ασαφείς, ανταυτόν θα έπρεπε να ακολουθήσουμε τις σαφέστερες κατευθυντηρίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Δεύτερη, η τροπολογία. Με αυτήν προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε ότι καλύπτονται και τα μεταποιημένα τρόφιμα στις οπολογίε 4, 5, 6 και 11 αναφερόμαστε στις πράξεις κάτω εξουσιοδότησης που θα έδιναν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να καθορίζει στοιχεία της πρότασης αυτής. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την τροπολογία 11 το πράττουμε αυτό να εξετάζει τις επιπτώσει που έχουν οι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά εξουσιοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να ακούσετε σχόλια των ε, σχεδόν. Είναι πραγματικά σπουδαίο. Και σε σχέση και όσον αφορά τη ε, Σύμφωνη Ελευθερών Εμπορίου ε, της Κύριε Φίσες, ο σκιώδης του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, ευχαριστώ για την κυρία Ντάρλινγκ για τα όσα ενδιαφέροντα μας εξήγησε. Πρόκειται για ένα σχέδιο κανονισμού που σχετίζεται με τα νέα τρόφιμα. Πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας. Ένας από τους στόχους είναι το πώς θα κατοχυρωθεί το καθεστώς που θα διέπει τα τρόφιμα που εισάγουμε από τις τρίτες ε, χώρες. Και βέβαια όλο και αυξάνει η ζήτηση και αυτό που μας ε, ενδιαφέρει να δούμε πώς θα διευκολυνθεί η εισαγωγή στην ευρωπαϊκή αγορά και την άλλη μεριά όμως δεν υπάρχει ασφάλεια όσον αφορά την ανάλωση αυτών των τροφίμων. Επίσης τώρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα όσον αφορά την κατοχήρωση των παραδοσιακών ε, τροφίμων της τρίτης χώρας και έτσι να υπάρχει ασφαλής χρήση και κατανοήση αυτών και έτσι θα, επίσης θα είναι ευκολότερη η πρόσβαση ε, ε, των ε, όσων εμπορεύονται από τις τρίτες χώρες αυτά τα τρόφιμα. Επίσης, όπως έχω πει στην συγκήτρια, να έχουμε κάποιες τροπολογίες για να δούμε ποιο, πώς, πώς θα φτάσουμε σε περισσότερη ασφάλεια για τα τρόφιμα. Θα πρέπει αυτό να ξεκαθαριστεί περισσότερο και να λάβουμε υπόψη ε, πώς θα υπάρχει ισορροπημένη διατροφή των Ευρωπαίων. Και αυτό θα πρέπει να έχει σαν κατοχήρωση, εύρος, να είναι συγκεκριμένο, όπου θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει από την ΕΦΣΑ κάποιες λεπτομέρειες, να μας πει ε, τις κατευθυντήριες γραμμές, τους κανόνες που ισχύουν τι, τι γίνεται. ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Πολύ καιρό τώρα θα θέλαμε να γίνει αυτή η ρύθμιση για τα νέα τρόφιμα και είναι σωστό το ότι τα κλωνοποιημένα εξαιρούνται. Δεν θα πρέπει όπως παρατηρήθηκε να έχουμε ρύθμιση που να αποτελεί φραγμό στο εμπόριο. και από που και σπού κάποια τρόφιμα τα οποία γνωρίζουν μαζί κατανάλωση εκτός Ευρώπη εμεί εδώ να τα έχουμε ε, περιορίσει. Επίση να γίνονται και ρυθμίσει τόσο ώστε να ωφεληθούν οι ΜΜΕ από τις εμπορικέ ροέ σε σχέση με αυτά τα τρόφιμα. Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει προ αυτή την κατεύθυνση και να υπάρχει τέτοιο νομικό καθεστώ, τόσο ώστε να είμαστε και εμεί βέβαια περισσότερο ανταγωνιστικοί. Και ταυτόχρονα να ωφεληθούν και χώρες εκείνες με ευκολότερη πρόοδο στην αγορά μας και ε, συμφωνούμε με τις τροπολογίες της Παρ' παρόλα αυτά έχουμε κάποιες ε, ε για το 11 εκεί που έχουμε αναβαθμισμένες αρμοδιότητες όσον αφορά την ΕΦΣΑ. Προσοχή τι, τι, τι ρυθμίσεις έχουμε σχετικά με την προσφυγή σε δικαστήριο, σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο, γιατί έτσι έχουμε κάποιο είδους ε, αυξημένη γραφειοκρατία και γενικότερα να δούμε πώς θα συνεχιστεί η λειτουργία της ΕΦΣΑ. Γενικότερα θα πρέπει πάντως επίσης να απλουστεύσουμε τις προηγούμενες διαδικασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει Ποιε είναι οι τροφές, ποια είναι τα τρόφιμα που καταναλώνονται από την πλειοψηφία του πληθυσμού στι τρίτε χώρε. Οπότε η ΕΦΣΑ συνεχίζει προ αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει και εμεί να δούμε μέχρι ποιου σημείο θα συνεργαστούμε. Για την άλλη, κύριε Σάντζη. Σας ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγήτρια για αυτό το προσχέδιο γνωμοδότησης. Πράγματι, είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί περαιτέρω, να είναι πιο σαφής ο ορισμός μάλλον των παραδοσιακών νέων τροφίμων. Υπάρχουν ε, τα παραδοσιακά νέα τρόφιμα τα οποία μπορεί να είναι πολύ γνωστά σε κάποιες τρίτες χώρες, αφενός και τα οποία καταναλώνονται μαζικά σε τρίτες χώρες στο παρελθόν, αλλά αφετέρου υπάρχουν και τα τρόφιμα που χρησιμοποιούν νανοηλικά. Εδώ είναι άλλο το ζήτημα. Τα θέματα της ε, διατροφής, της ασφάλειας των τροφίμων είναι κρίσιμες σημασίας. Αναφέρατε και εσείς τις διαπραγματεύσεις για την TTIP. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο ευρωπαϊκό, το οποίο θα διασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη και στο μέλλον και πρέπει να εξασφαλίσουμε, να διασφαλίσουμε το μέλλον, με συγχωρείτε μάλλον την ασφάλεια των καταναλωτών βραχυπρόθεσμα αλλά και, και μακροπρόθεσμα. Θέλω να αναφερθώ σε κάποια κύρια σημεία. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα της αρχής της προφύλαξης, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται και να συνεχίσει να εφαρμόζεται και πρέπει να το επαναλάβουμε αυτό και αφορά και τα νέα τρόφιμα η αρχή της προφύλαξης θα πρέπει να συνεχίσει να διέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο στον τομέα αυτών. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει ε, λασιμότητα, απόλυτη λασιμότητα όσον αφορά τα συστατικά στοιχεία των τροφίμων αυτών. Και οι πληροφορίες σχετικές θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και κατανοητές από οποιονδήποτε επιθυμεί. Τρίτον, βεβαίως και θα πρέπει να να μην συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία τα προϊόντα από κλόνους. Είμαστε εν αναμονή ενό νέου κειμένου για το ζήτημα αυτό. Και τέταρτον θέμα, πιστεύω ότι θα, έχει, θα ήταν σκόπιμο να σκεφτούμε με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόντεξ αλιμεντάριος, εκεί όπου πραγματικά λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων διεθνώς και πώς μπορούμε να προωθήσουμε ένα ε, πλαίσιο ασφάλειας τροφίμων κοινό για όλες τις χώρες μέλη του κόντεξ. Πρέπει να ε, ενισχύσουμε τη θέση μας στον κόντεξ, πιστεύω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Μίνερ. Ik kan instemmen met de ευχαριστώ. Σύμφωνο με τις ε, προτάσεις και τις τροπολογίες που προτείνει η κυρία Ντάρλινγκ, το σημείο εκκίνησης και το πιο σημαντικό στοιχείο πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων. Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πώς θα εξασφαλιστεί αυτή. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση, τη λογοδοσία, να εξασφαλίζει ότι οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση θα είναι και περιορισμένες και οι απολύτως απαραίτητες. Η προέλευση, η χνηλασιμότητα είναι θέματα σημαντικά. Υπάρχουν επίσης, υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ αυτής της συγκεκριμένης πρότασης και της υπόλοιπης συζήτηση που γίνεται για παράδειγμα για την TTIP. κύριος Γιάννικ. Ναι, ευχαριστώ. Όπως είπε και η Μαρή, ξεκινάμε με το κείμενο αυτό μια μεγάλη και δύσκολη συζήτηση για το ζήτημα των νέων τροφίμων και καλό είναι να θυμούμαστε ότι το ζήτημα που διακυβεύεται δεν είναι μόνο τα κλωνοποιημένα τρόφιμα, τα, συγγνώμη, τα τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα, τα οποία προφανώς και πρέπει να απογορεύσουμε, αλλά επίσης και τα μεταποιημένα τρόφιμα από, από κλώνους. Όσον αφορά τώρα τα παραδοσιακά νέα τρόφιμα. Το δίλημα εδώ είναι πως μπορούμε και, να διευκολύνουμε το εμπόριο και να αγγιηθούμε την ασφάλεια. Θα έλεγα ότι εμείς ε, υποστηρίζουμε περισσότερο την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή τη μελέτη του ιστορικού, της χρήσης, της κατανάλωσης αυτών των τροφίμων σε ένα βάθος χρόνου 25 ετών κτλ. Αντιθέτως, μια προσέγγιση η οποία θα έδινε μεγαλύτερο ρόλο στην ΕΦΣΑ στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλεια των Τροφίμων, δεδομένου ότι οι απαραίτητε μεταρρυθμίσει στην ΕΦΣΑ δεν έγιναν. Θα μπορούσαν να οδηγήσουν το να εγκριθούν ως παραδοσιακά νέα τρόφιμα, ε, τρόφιμα τα οποία στην πραγματικότητα είναι μεταλλαγμένα. Το άλλο θέμα το οποίο μας ανησυχεί είναι τα μεταποιημένα τρόφιμα. Να μην ονομαστιστούν μεταποιημένα τρόφιμα ως παραδοσιακά, δεδομένου ότι τα μεταποιημένα, στα μεταποιημένα τρόφιμα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθεί νέα υλικά. Αυτό μας προβληματίζει για παράδειγμα, χρήση νάνο υλικών σε ένα τρόφιμο ε, το οποίο θα ονομαστεί μεταποιημένο παραδοσιακό τρόφιμο. Αυτό ο κυκλικό ορισμό μας προβληματίζει, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία στα οποία θέλουμε εμεί να επιμένουμε. Ευχαριστούμε. Ευρώπη των Ελευθεριών και των Δημοκρατιών βλέπω να μην ζητάει το λόγο. Θέλει κανείς άλλο το λόγο εκ των συναδέλφων. Όχι. Η Επιτροπή τότε. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο που έχω στον καταλογό μου, Σαντάλ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συγητή τους και τους συγητές επίσης, γιατί ήταν πάρα πολύ ε, ενδιαφέροντα τα όσα είπαν. Είμαστε θετικοί όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για τα νέα τρόφιμα Απλώς, πράγμα είναι όταν ε, είχε υποβληθεί πρόταση αρχικά, είχαμε και δύο προτάσεις για την κλωνοποίηση. Ε, είχε υποβληθεί σχετική πρόταση σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και βεβαίω η πρόθεσή μας ήταν ε, όσο δεν εγκρίνονται αυτά τα κείμενα τότε να καλυφθεί η υπόθεση των κλωνοποιημένων από το κείμενο για τα νέα τρόφιμα για να μην υπάρχει κενό στην νομοθεσία. Επίσης, συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση, ε, βοηθά την καινοτομία στην Ευρώπη, θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να έχουν πρόταση στην χώρα, ε, γιατί θα διευκολυνθούν οι αδειοδοτήσεις. Επίσης είναι σημαντικό το ότι η νομοθεσία θα βοηθήσει για περισσότερη διατροφική ασφάλεια, θα προστατευτούν οι καταναλωτές και τώρα όσον αφορά την βασική αρχή για τα τρόφιμα της τρίτες χώρες βεβαίως και θα πρέπει να υπάρχουν τα ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας όπως και τα τρόφιμα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα και όπως τονίστηκε από συναδέλφους το πιο σωστό είναι ε, αφού έχουμε κάποια τρόφιμα ε, θεωρούνται παραδοσιακά αυτά τα οποία με ασφάλεια καταναλώνονται στις τρίτες χώρες δεν είναι παραδοσιακά για την ε, ε, Ευρώπη. Το κριτήριο είναι το αν στο, στο τρόπο διατροφής αυτά είναι που επομένως παγίως χρησιμοποιούμενα χρειάζεται και για αυτά επομένως με το δίκτυο ασφαλείας αυτή η διαδικασία κοινοποίηση και αν υπάρχει ένσταση από τα κράτη-μέλη τότε συγκεκριμένο τρόφιμο ε, δεν θα καλύπτεται από αυτή την απλή κοινοποίηση και θα πρέπει να περάσει από πιο πολύπλοκη διαδικασία. Και δικαιολογείται η σύντομη διαδικασία εάν επομένω για, για 25 χρόνια ή πάνω από μια γενιά έχει καταναλωθεί αυτό το τρόφιμο και έτσι. Και σας παραπέμπω στις ε, συζητήσεις τη συνδιαλλαγής για τις προηγούμενε προτάσει και έτσι τέλο πάντων έχουν μια ευκαιρία οι τρίτε χώρε και είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί στην οδηγία ε, η έννοια της ε, παραδοσιακής ε, διατροφής ούτω ώστε να ωφεληθούν οι τρίτες χώρες και να μπορέσουν για κάποια τρόφιμα να έχουν την σύντομη διαδικασία της κοινοποίησης. Να δούμε τι θα γίνει και με την πρωτογενή παραγωγή όπως κάποια χυμή φρούτων, όπως κάποια του τροφίμων τα διατροφή, συγγνώμη, τα, τα οποία ποτέ δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι είδο παραδοσιακή διατροφής, γιατί πάντα είναι κάτι το κατεξαίρεση χορηγούμενο, λαμβανόμενο. Και θα πρέπει πάντοτε να έχουμε κατανόηση, θα πρέπει για τι τρει χώρε να ισχύουν οι ίδιες προγραφέ ε, ασφαλείας και θα πρέπει επομένω ό,τι η διαδικασία ισχύει να ισχύει για όλους, και την Ευρώπη και τις τρίτες χώρες. Και, εν πάση να τίθεται σε, να τίθεται σε εμπορία ασφαλή τρόφιμα στην Ευρώπη. Υπάρχει νομοθεσία και ισχύει όπου υπάρχει αβεβαιότητα για το αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος Οπότε ισχύει η αρχή της ε, επιφύλαξης. Και αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα για αυτό το σκοπό θα συνεχίσουν να ισχύουν. Στην πρότασή μας, αλλά και στην πρόταση που συζητήθηκε στη συνδιαλλαγή, πρόθεση μας δηλαδή, δεν ήταν το να διευρύνουμε το πεδίο μαγείς αυτού του κειμένου. Θέλαμε απλώς το υπάρχον κείμενο να διευκρινιστεί. Άρα εδώ επιδέχεται βελτιώσει τεχνικό επίπεδο το κείμενο, ούτω ώστε να βελτιωθεί ο ορισμό να εξασφαλίσουμε ότι το πεδίο εφαρμογή για όλους θα είναι κάτι το συγκεκριμένο, για όλους και, και τους εμπορευόμενους και τις ε, κυβερνήσεις, ούτως ώστε να υπάρχουν οι δέοντες έλεγχοι όσον πρέπει την αναθεώρηση μετά την πενταετία, όπως είπε η συγκήτρια, θα προτιμούσαμε αυτή η αναθεώρηση να γίνει στα πλαίσια της αξιολόγησης της ε, Κομισιόν για το, γενικότερα για τον αποτελεσματικό της νομοθεσίας. Να δούμε δηλαδή εάν καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει με αυτό το νομοθέτημα. Και δεν ξέρω μήπως αυτή η πενταετία είναι κάτι το σύντομο, μήπως θα πρέπει να γίνει αυτό λίγο αργότερα για να δούμε εάν μπορούμε να έχουμε μια αποτελεσματική ανάλυση για τις επιπτώσεις του νομοθετήματος. Όσον αφορά τώρα την κατεξοδότηση πράξη και την εφαρμογή αυτής θα πρέπει να δούμε αν οι όργοι προποθέσει που ισχύουν πληρούνται. Εν κατακλείδη, ευχαριστούμε την εισηγήτρια και τους κοιόδους εισηγητές για την ανταπόκρισή τους στην θετική και ελπίζουμε το συντομότερο δυνατόν να εγκρίνεται την πρότασή μας γιατί είμαστε σίγουροι ότι αυτή η συντομότερη διαδικασία έγκρισης θα ωφελήσει όλους και στην Ευρώπη και στις τρίτες χώρες και επίσης θα βοηθήσει για την διατροφική ασφάλεια. Δίνω τον λόγο στην εισηγητρία μας. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και για το γεγονό ότι υποστηρίζουν σε γενικές γραμμές την προσέγγιση που έχω ακολουθήσει. Δύο-τρία πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, ο ρόλος της ΕΦΣΑ νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν περισσότερο οι κατευθυντήριες ε, οδηγίες της ΕΦΣΑ, γιατί αυτό θα μας δώσει επίσης τη δυνατότητα να, να ξεκινήσουμε ένα διάλογο με τους διεθνείς οργανισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων. Δεύτερον, για το σχόλιο του κυρίου Γιάννη, για τα 25 έτη εδώ κρατήσαμε την αναφορά στα 25 χρόνια στο κείμενο. Το ζήτημα είναι άλλο. Το ζήτημα είναι ότι γίνεται μια αναφορά στην παραδοσιακή διατροφή ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού με αυτής της τρίτης χώρας. Και αυτό είναι ασαφές. Ο ορισμός θα έπρεπε να είναι πιο συγκεκριμένος. Και βεβαίως να το συζητήσουμε με την Επιτροπή, αν ίσως να μας πείσουν ότι ο ορισμός που προτείνουν είναι καλύτερος. Ε, πάντως εμείς θα θέλαμε οι ορισμοί να γίνουν πιο συγκεκριμένοι και σαφείς. Τώρα, ε, στο προσεχέ μέλλον θα σα παρουσιάσω τι δύο γνωμοδοτήσεις, προσχέδια γνωμοδοτήσεων για την κλωνοποίηση. Τότε θα κάνουμε τη σχετική συζήτηση για την κλωνοποίηση. Σα ευχαριστώ για τα σχόλιά σα Ευχαριστώ να συναντηθώ και με του κοιόδη συζητητέ για να συζητήσουμε το θέμα τι επόμενε μέρε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών η 10 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι. όπου θα συζητηθούν και πάλι στις 5 και 6 Νοεμβρίου οι τροπολογίες για να ψηφίσουμε μάλλον στις 6. Θέλω να επισημάνω ότι η αρμόδια καθήλυν Επιτροπή, Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει σήμερα μία ακρόαση προγραμματίσει για τις 12 και 4 και άρα Ίσως έχετε τη δυνατότητα να αποκομίσετε ε, ειδικότερε και εις βάθος πληροφορίες. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτό το θέμα και προχωρώ στο επόμενο, στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι το υπαριθμό 11 και το θέμα των διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ιαπωνίας για το εμπόριο. Έχουμε τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή κύριο Μάουρο Περτιτσόνη εδώ από τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικού Εμπορίου και τον παρακαλώ να λάβει το λόγο. Πριν όμως από αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Πέντρο Σίλβια Περέρα που είναι ο μόνιμος ε, εισηγητής για τα θέματα των σχέσεων με την Ιαπωνία. Τον καλό λοιπόν τον κύριο Περέιρα πριν λάβει το λόγο η Επιτροπή να μας κάνει μία εισήγηση για το θέμα αυτό. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και επιτρέψτε μου καταρχάς να πω ότι με τιμά το ότι έλαβα τον, ε, ανέλαβα καθήκοντα μόνη μου εισήγητη για τη σχέση με την Ιαπωνία Σα ευχαριστώ πολύ. Με χαρά θα συνεργαστώ μαζί σας, όπως και με την προηγούμενη σύνθεση της Επιτροπής πριν τις εκλογές, για την διερεύνηση των σχέσεων. Εάν ήταν η πρώτη εμπορική συμφωνία στην οποία έδωσε σύμφωνη γνώμη το Κοινοβούλιο αυτή της Κορέας, των σχέσεων με την Κορέα, η Ιαπωνία ήταν η πρώτη διαπραγμάτευση που ξεκίνησε υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του εξετάζει πολύ προσεκτικά από τα πρώτα βήματα αυτή την διαδικασία η οποία οδηγεί στη συνέχεια στην έναρξη των συνομιλιών. Έχουμε αποστείλει αντιπροσωπεία στην Ιαπωνία σε ένα πρώιμο στάδιο. Είχαμε εκεί, είχε εκεί η αντιπροσωπεία αυτή επαφές όχι μόνο με Ευρωπαίους ε, φορείς αλλά και με κύριους παράγοντες από πλευράς Ιαπωνικής σε πρώιμο στάδιο. Στη συνέχεια προχώρησε στην σύνταξη ε, της εντολής για το... Ε, θα έπρεπε να προχωρήσει στη σύνταξη εντολής στο Συμβούλιο αλλά το Κοινοβούλιο παρενέβη τόσο από το Συμβούλιο να επιφυλαχθεί ακόμα μέχρι ότου το Κοινοβούλιο ορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπραγμάτευση και με την πίεση, πίεση αυτή και το σημαντικό αυτό βήμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει μια νέα διοργανική πρακτική που έκτοτε εφαρμόζεται στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο με τρίτες χώρες. Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε το Συμβούλιο προσεκτικά μελέτησε τις θέσεις του Κοινοβουλίου με σαφή ένδειξη την ε, ετήσια επισκόπηση των συνομιλιών που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2014 και όπου καταγράφονται και τα αιτήματα του Κοινοβουλίου όπως είχαν εκφραστεί με τα ψηφίσματά μας. Επιπλέον το Κοινοβούλιο παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την, ε, τις θέσεις των εμπλεκομένων ευρωπαϊκών φορέων, επιχειρήσεων και τη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις. Αντιλαμβανόμεθα ότι έχουν εκφραστεί σημαντικές ανησυχίες ως προς την ε, ε, θέση και την κατάσταση της ε, αυτοκινητοβιομηχανίας που αντιμετωπίζει μη δασμολογικούς φραγμούς στην Ιαπωνία. Ένα άλλο ζήτημα ήταν αυτό των δημοσίων προμηθειών και το γεγονός ότι ε, αποκλείονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τον κλάδο των Ιαπωνικών συνδυροδρόμων. Επίσης με μεγάλη προσοχή παρακολουθήσαμε τις τοποθετήσεις των φορέων εκείνων που έχουν εκφράσει τη δυνατότητα για πρόσβαση ε, που έχουν εκφράσει την ανάγκη για μια καλή δυνατότητα για πρόσβαση στην ιαπωνική ε, αγορά καθώς και των ιαπωνικών επιχειρήσεων που θέλουν πρόσβαση και δραστηριότητες στην ευρωπαϊκή αγορά. Τώρα παρακαλώ τον, ε, να ακούσουμε τον κύριο Πετριτσάνη, γιατί περιμένουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσω τις θέσεις του και πάνω απ' όλα ή πρώτα απ' όλα οποιαδήποτε ενημέρωση έχει να μας δώσει για το τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων, τις προσδοκίες για τον προσεχή γύρο που αναμένεται στο τέλος του μήνα και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Ιαπωνίας με το φύλλο πορείας, οδικό χάρτη και το στόχο του εκμηδενισμού των μη δασμολογικών φραγμών. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πετροτσάνη πώς βλέπει την ε, ισχύουσα κατάσταση σε σχέση με την υλοποίηση του φύλου πορείας ως προς τους και τις αστικές μεταφορές. Τι είδους δεσμεύσεις έχετε λάβει από πλευρά Ιαπωνικής πως Ευρωπαίοι φορείς και επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση στην Ιαπωνική αγορά ε, και τις δημόσιες προμήθειες της Ιαπωνίας γιατί έχουν εμφανιστεί σοβαρές ανησυχίες πως η ρήτρα προστασίας όπως υφίσταται αυτή τη στιγμή θα εξακολουθήσει να αποτελεί πρόσκομα για την ε, συμμετοχή στο σχέδιο αυτό ε, διαφάνειας στην αγορά της Ιαπωνίας. Επίσης υπάρχει το ζήτημα των αυτοκινήτων όπως ονομάζεται cars, Υπάρχει δηλαδή η απαγόρευση για, για πώληση ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στην Ιαπωνική αγορά. Υπάρχει το ζήτημα των ε, ενδείξεων γεωγραφικής προελεύσεως, όπου ελπίζουμε να δούμε μια κάποια πρόοδο. Και επίσης αν οι δασμολογικές, οι προσφορές σας προς τα δασμολογικά που έχουν ε, ε, ανταλλαγή είναι ικανοποιητικές ή τι είδους φιλοδοξίες έχετε ως προς αυτές. Ασφαλώς μας ενδιαφέρει η πρόοδος και στο χώρο των ε, γεωργικών ε, προϊόντων και τροφίμων. Θέλουμε να δούμε τις θέσεις σας και τις προσδοκίες σας. το κεφάλαιο για την αηφόρο ανάπτυξη επίσης μας ενδιαφέρει πολύ και θέλουμε να δούμε εάν υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πατριτσόν έχει το λόγο. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ιδιαίτερα ευτυχίες που μου δίνετε τη δυνατότητα να απευθυνθώ στην ΙΝΤΑ για να σας ενημερώσω ε, για την σχέση μας με την Ιαπωνία. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Επιτροπή σας μετά τις ευρωεκλογέ. Θα σας ενημερώσω σύντομα, σύντομα συνοπτικά τι έχει γίνει μέχρι τώρα που βρισκόμαστε και μετά θα προσπαθήσω να απαντήσω ε, στα ερωτήματα του κυρίου Περέιρα. Αυτή η διαπραγμάτευση είναι μία από τις πλέον σημαντικές που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν αναλογιστούμε τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει, τι θετικές επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι όμως και μία από τις πιο περίπλοκες ε, διαπραγματεύσεις θα έλεγα περισσότερο από την συμφωνία με τον Καναδά και συγκρίσιμα περίπλοκη με την TTIP, με τις ε, συγγνώμη, εμπορικές τη της ΗΠΑ. Η Ιαπωνία είναι μια χώρα με αναπτυγμένη οικονομία, περίπλοκα συστήματα. Ο λόγος ο βασικός που μας έχει δοθεί η δυνατότητα να διαπραγματευτούμε με τους Ιάπωνες είναι επειδή εκείνοι αποφάσισαν ότι θέλουν να αλλάξουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ασκούν την οικονομική τους πολιτική. Έχουν ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων το οποίο μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούμε με την τρέχουσα Ιαπωνική κυβέρνηση η οποία έχει και την εντολή και την πολιτική βούληση και το σχέδιο για να ελοποιήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ε, θα γνωρίζετε ότι οι κυβερνήσεις στην Ιαπωνία ε, δεν ήταν και τόσο σταθερές τα τελευταία χρόνια και δεν είχαν γι' αυτό το λόγο τη δυνατότητα να λαμβάνουν φιλόδοξα προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Έχουμε λοιπόν τώρα μία ευκαιρία. Ε, υπάρχει το ζήτημα των αυτοκινήτων, των δασμών και γενικότερα. Το σημαντικότερο θέμα για την Ιαπωνία αναφέρεται ως η άρση των ε, περιορισμών εξαιτία των δασμών, αλλά στην πραγματικότητα αυτά που συζητάμε είναι πώς θα προσεγγίσουμε ε, την Ιαπωνία, πώς και η Ιαπωνία θα έρθει και πιο κοντά σε εμά στον τομέα του ρυθμιστικού πλαισίου. Το καλό είναι ότι η Ιαπωνία συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε γενικές γραμμές όσον αφορά τα πρότυπα τα περιφερειακά. Διαφωνούμε μαζί τους συχνά στον τρόπο με τον οποίο τα περιφερειακά πρότυπα πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο και αυτό είναι το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων μαζί του, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τις, ε, τα διεθνή πρότυπα και τα περιφερειακά πρότυπα συμφωνούμε μαζί του. Υπάρχει λοιπόν μια καλή ευκαιρία να συγκλίνουμε. Έρχομαι τώρα στα ερωτήματα του κύριου Περέιρα, τα πιο συγκεκριμένα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις. Θα έλεγα ότι ε, ήταν μια από τις πολύ καλά προετοιμασμένες διαπραγματεύσεις μας. Ε, η διαδικασία προετοιμασίας ξεκίνησε πριν τέσσερα χρόνια και ήταν η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγε μια πλήρη αξιολόγηση αντικτύπου πριν ξεκινήσει την διαπραγμάτευση. Επίση, έγιναν συζητήσει ε, διοξοδικές και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έντονε συζητήσει και στο Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά. συνεχίζει να υπάρχει ένα μάλλον υπήρχε η εκκρεμότητα, η αμφιβολία το κατά πόσον η, η Ιαπωνία ε, ήταν αποφασισμένη να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις του συστήματος των δασμών, το οποίο οδήγησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, δημιουργήσει μια ρήτρα μετα... Ε, αναθεώρησης. Έγινε αυτή η αναθεώρηση που διήρκησε ένα χρόνο. Όσον αφορά τον περιορισμό των φραγμών από τους δασμούς στον τομέα των αυτοκινήτων, η Ιαπωνία επιθυμεί να ακολουθήσουμε τα διεθνή πρότυπα, να συμφωνήσουμε σε ένα σχέδιο για την Ιαπωνία, με το πρόγραμμα εργασιών με το οποίο η Ιαπωνία θα εφαρμόσει το διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο με τον ίδιο τρόπο που το έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το λεγόμενο cold plating, δηλαδή η υιοθέτηση ενός διεθνούς προτύπου, αλλά με μια μικρή προστίκη, η οποία στην πραγματικότητα δημιουργεί φραγμούς σε εταιρείε από το εξωτερικό να δραστηριοποιηθούν στην αγορά σου. Πρότεινε λοιπόν η Ιαπωνία ένα πρώτο πακέτο μεταρρυθμίσεων. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τα Ιαπωνικά Υπουργεία. Έχουν ήδη εγκρίνει κάποιες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Συμφωνούμε επίσης μαζί τους στο ρυθμιστικό πλαίσιο ήταν ε, παροχημένο και θα συνεργαστούμε έτσι ώστε να προκαλέσουμε και μια αναθεώρηση του ίδιου του ρυθμιστικού πλαισίου στο επίπεδο της UNEC. Το επόμενο ζήτημα ήταν τα προσθέτα τροφίμων. Έχουμε επιτελούς συμφωνήσει σε έναν κατάλογο πρόσθετων τροφίμων αυτός ο κατάλογος συζητιόταν επί χρόνια παλαιότερα και υπάρχει και το ε, γνωστό ε, σχέδιο για τους σιδηροδρόμους. Στο πλαίσιο των συζητήσεων για τις δημόσιες συμβάσεις είχε υπάρξει μια ε, δέσμευση η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ρήτα ασφαλείας που δίνει τη δυνατότητα στην Ιαπωνία, έδινε τη δυνατότητα μάλλον στην Ιαπωνία να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας. Χρειάζεται λοιπόν συζήτηση για να διευκρινιστεί ποιε είναι ακριβώ αυτέ οι απαιτήσει ασφαλείας, πώ θα εφαρμόζεται αυτή η ρήτρα ασφαλεία και ότι οι ευρωπαϊκοί οικονομικοί φορεί θα έχουν τη δυνατότητα να αποδεικνύουν στα στι Ιαπωνικέ αρχέ ότι πληρούν τι εξαιρετικά υψηλέ Ιαπωνικέ απαιτήσει για την ασφάλεια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι γνωστέ αυτέ οι απαιτήσει ασφαλεία. Αν απλώ υπάρχει αυτή η ρήτρα χωρί να είναι σαφέ ποιε απαιτήσει θα πρέπει να πληρούνται, οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει ούτε καν θα προσπαθήσουν να εισαγούν τι δραστηριότητε του εκεί. Πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί σε ποιε περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να ενεργοποιηθεί αυτή η ρήτρα ασφαλεία. Υπάρχουν επίσης εθελοντικοί κανόνες συμπεριφοράς, ε, λειτουργίας μάλλον, των τριών ιδιωτικοποιημένων πλέον ε, ε, ε εταιριών ε, σιδηροδρόμων Έχουμε και εμεί έναν ευρωπαϊκό και κώδικα εθελοντικό που έχει πολύ παρόμοιε προβλέψει. Το αποτέλεσμα όμω αυτό δεν μα ικανοποιεί πλήρω γιατί δεν λύνει το πρόβλημα τη πρόσβαση στην αγορά. Για παράδειγμα, το γεγονό ότι η ρήτρα ασφαλεία μπορεί να ε, εφαρμοστεί σε πολλά και διάφορα ε, είδη τεχνικού εξοπλισμού. Πρέπει λοιπόν να λυθεί αυτό το ζήτημα αυτή της, της ασάφειας που υπάρχει με τη ρήτρα ασφαλείας, σε ποιο είδος εξοπλισμού εφαρμόζεται, σε ποιες περιπτώσεις. Και το ζήτημα γενικότερα της πρόσβασης αγορά θα συνεχίσει να επανέρχεται στη διαπραγμάτευση. Η Ιαπωνική πλευρά ε, ολοκλήρωσε αυτά που έπρεπε να ολοκληρώσει στο πλαίσιο του μονοετούς προγράμματος αναθεώρησης. Αυτή τη στιγμή συζητείται το θέμα στο Συμβούλιο έτσι ώστε και εμείς να εκπληρώσουμε τις ε, δικές μας υποχρεώσεις. Το ζήτημα είναι περίπλοκο και τεχνικό. Εμείς ποτέ δεν είχαμε δεχτεί ότι αυτές οι τρεις εταιρείες ε, θα εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις της GPA. Εάν η Ιαπωνική πλευρά κάνει παραχωρήσεις στο ζήτημα της ρήτρα ασφαλείας, θα μπορούσαμε να δεχθούμε τη διαγραφή τους, γιατί έτσι και λέω πλέον είναι ιδιωτικές εταιρείε και εφαρμόζονται γενικώ ο για τις ιδιωτικές εταιρείε, δεν τίθεται θέμα. Η συνεργασία με τα Υπουργεία, ιδίω εκείνα που ασχολούνται με τεχνικά θέματα, είναι πολύ καλή. Και αυτό μας ε, δημιουργεί την πεποίθηση ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση ε, εγκαίρως, γρήγορα, χωρίς να έχουμε κάποια συγκεκριμένη προθεσμία. Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός Άμπε έχει ε, προτείνει τον Ιούλιο του 2015 ως ε, την προθεσμία, δεδομένου ότι οι εκλογές στην Ιαπωνία θα γίνουν τον Ιούλιο του 2016. Είναι φιλόδοξος στόχος, αλλά πετύχω, ε, πιστεύω εφικτός. ότι είμαστε... Ε, έχουμε την πεποίθηση ότι μπορεί να γίνει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προσπαθήσουμε. Έχουμε πολύ καλή σχέση με την Ιαπωνία, αλλά η διαπραγμάτευση είναι δύσκολη. Τα τελευταία 40 χρόνια είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη έχει καλέ σχέσει με, με του Ιάπωνε, αλλά οι διαπραγματεύσει δεν είναι απλέ. και ε, έχουμε στη διάθεσή μας ένα χρόνο και κάτι αρκεί αλλά δεν θα έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε λάθη και να επανέλθουμε σε θέματα πολλές φορές. Τώρα, έρχομαι στα ερωτήματα της συγκεκριμένα του κ. Περέιρα. Ανέφερθηκα ήδη σε κάποια από αυτά τα θέματα. Το πρώτο ζήτημα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ήταν τα πρότυπα για τα οχήματα της UNEC. Οι εξαγωγέ ε, αυτοκινήτων από την Ιαπωνία έχουν αυξηθεί. Όμως, κυρίως αυτά που εισάγονται είναι αυτοκίνητα πολυτελείας μάλλον εξάγονται από την Ευρώπη προς την Ιαπωνία είναι κυρίως ε, γνωστές μάρκες και πολυτελή αυτοκίνητα. Δεν πολλούμε ας πούμε, πολλά Fiat Punto, τα Cinquecento όμως έχουν ισχυρές πωλήσει στην Ιαπωνία. Αυτό σημαίνει ότι είναι συγκεκριμένα είδη αυτοκινήτων τα οποία έχουν κερδίσει τους Ιαπωνές καταναλωτές, όμως εμείς δεν θέλαμε να αυξήσουμε συνολικά τις πωλήσει εκείνων των αυτοκινήτων που έχουν υψηλές πωλήσει στην Ευρώπη αλλά όχι στην Ιαπωνία. Και για αυτά τα αυτοκίνητα το θέμα των προτύπων των τεχνικών είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί το ζήτημα τα ιαπωνικά αυτοκίνητα δεν είναι μόνο ότι είναι τεχνικά άρτια αλλά είναι και φτηνά. Επομένω, εάν η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία θέλει να κερδίσει σε μια αγορά όπου το περιθώριο κέρδου είναι σφιχτό, είναι ε, περιορισμένο, το ζήτημα των τεχνικών προτύπων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μέχρι πρόσφατα δεν είχε εμφανιστεί το ζήτημα των key cars να είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μέχρι το 30% της αγοράς αυτοκινήτων στην Ιαπωνία ε, έχει σχέση με αυτό το είδος αυτοκινήτου, ωστόσο λίγες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη παράγουν μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα Ιαπωνικά. Φαντάζομαι λοιπόν ότι εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούσε να συμφωνήσει σε κάποια ε, ευρωπαϊκούς ε, δασμούς για τα αυτοκίνητα αυτά θα είχαμε τις ενστάσεις των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά πάσα πιθανότητα. Εάν δεν αλλάξει λοιπόν το φορολογικό καθεστώς για τα αυτοκίνητα στην Ιαπωνία έχει ξεκινήσει μια διαδικασία μάλλον αναθεώρησης του φορολογικού καθεστώτος των αυτοκινήτων. Ανάλογα με το πώς εκείνη θα εξελιχθεί, φαντάζομαι ότι θα μεταβάλει και τη στάση της στο ζήτημα των δασμών. Μέχρι τώρα προσπαθούσαν να προωθήσουν τα μικρά αυτοκίνητα ε, με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μηχανής το μέγεθος του αυτοκινήτου και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, ε, η ευρωπαϊκή Βιομηχανία γνωρίζει το θέμα αυτό. Γεωγραφική ένδειξη. Αυτό είναι κάτι το πιο δύσκολο. Παραδοσιακά δείχνει κατανόηση για το δικό μας ε, νομικό καθεστώς η Ιαπωνία και επίσης βρισκόμαστε στι συνομιλίες ε, και εκείνη με τις Ηνωμένες οι Ιαπωνοί θέλουν να υπάρξει κάποια ρύθμιση για το σήμα ευρεσιτεχνίας οπότε κάνουν κάποιες βελτιώσεις αλλά ακόμα δεν είμαστε ικανομένοι πλήρως συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις και αυτό το οποίο θέλουμε βέβαια είναι να πετύχουμε κάτι σαν αυτό που πετύχαμε με τον Καναδά ε, βέβαια δεν είναι εύκολο αυτό, το ξέρουν οι Ιαπωνέζοι και στις διαπραγματεύσεις ε, το χρησιμοποιούν αυτό ε, και άλλα νομοθετούν στο ιστορικό της χώρας και άλλα λένε στις διαπραγματεύσεις με εμά. Τώρα, όσον αφορά τους δασμούς, όσον αφορά τα αγροδιατροφικά, τα είπαμε, έχουμε κάποιες μελέτες επιπτώσεων και βέβαια αυτός ο κλάδος θα είναι ο πρώτος μακράν που θα ωφεληθεί από την ε, εμπορική συμφωνία. Αυτό που καταρχήν προσφέρουν ε, οι Ιαπωνέζοι από εμά είναι αποδεκτό. Καλύτερη πρόσφατα θα μπορούσε να γίνει και θα πρέπει να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Είναι σαφές ότι η Ιαπωνία θέλει εμείς για τα αυτοκίνητα και για άλλα βέστα προϊόντα να μειώσουμε τους δασμούς αλλά και πρέπει θα το κάνουμε αυτό αν θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στην αγορά τους ε, για κάθε προϊόν. ο πρόεδρε, ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ο πρόεδρος. Συνάδελφοι, να είστε παρακαλώ σύντομοι, ακριβείς στις ερωτήσεις σας, αλλιώς δεν θα μείνει χρόνος για να συζητήσουμε το επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης. Κύριος βαλεσα για το ΕΛΚ. Σύντομη ερώτηση. Είπαμε ότι η εφαρμογή ε, του, του πακέτου του ενός έτους για τα ε, θα ε, εξαρτιόταν από το αν θα συμφωνήσουν οι, Ιαπωνέζοι για τις ρυθμίσεις που υπάρχουν όσον αφορά να κάνουν δηλαδή στην, αγορά τους αυτά τα οποία τους έχει πει να κάνουν ε, ο ΠΟΕ και, για το, και γενικά για το προτιμησιακό καθεστώς που ισχύει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ε, την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ακόμη όμως δεν είναι σαφές ότι μπορούμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει διαφάνεια για τις σχετικές εταιρείε. Ακόμη υπάρχουν δυσμενείς διακρίσεις όσον αφορά τους διαγωνισμούς ε, των προμηθειών. Δεύτερη ερώτηση. Δεν αποδεικνύεται έτσι το πόσο δύσκολο είναι το να μπορέσουμε να έχουμε αυτή του τη, μόχλευση. Και δεν μπορούμε έτσι να παρακάμψουμε τους περιορισμούς που βάζει η Ιαπωνία όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά τη. Επόμενο ο κύριο Ζαχραντή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα περισσότερα τα κάλυψε ο εισηγητή. Είπε όλα τα σχετικά με τους κρατικούς διαγωνισμούς και για την κατάρριξη των μη δεσμολογικών φραγμών Οπότε έχω δύο δευτερόλεπτα πράγματα να ρωτήσω. Πρώτα πρώτα. Δεν κατάλαβα αν κατάλαβα σωστά τα όσα ελέγχθησαν περί φορολόγησης. Μας είπατε τι γίνεται με αυτά τα μικρά αυτοκίνητα, τα ευρωπαϊκά. Μήπως μπορείτε να ε, μας τα, το αναλύσετε καλύτερα. Ε, δεύτερον, πώς έχει η κατάσταση για τις χρηματοοικονομικές και νομικές υπηρεσίες όσον αφορά δηλαδή Ευρωπαίους που θέλουν να πάρουν τις υπηρεσίες στην Ιαπωνική αγορά κάτι αναφέρθηκε αλλά μπορείτε και αυτό κάπως να το εξηγήσετε περισσότερο Μαρίκε Μαρίκε Πώς να μας δίνει ευκαιρία να συζητήσουμε τις διαπραγματεύσεις μας με την Ιαπωνία. Είπαμε πολλά για τους κρατικούς διαγωνισμούς, τις προμήθειες και εγώ θέλω να ακούσω περισσότερα και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για ένα πάρα πολύ καυτό θέμα. Το ISTS, δηλαδή η Αυστραλία και η Ιαπωνία έκλεισαν μια εμπορική συμφωνία χωρίς το ISTS. Να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορεί τι συζητείτε σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια. Τι γίνεται με την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Έπαιξε κάποιο ρόλο η τραγωδία της Φουκουσίμα. Επίσης, τι γίνεται με τις ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα παγώσουμε τις συμφωνίες ε, εάν κάτι δεν γίνει με την, ε, ε, με την θανατική ποινή που ισχύει στην Ιαπωνία. Να ευχαριστήσω για το όσα ακούσαμε και έχω τις εξής τρεις ερωτήσεις. Κάνουμε τις διαπραγματεύσεις σε ένα πλαίσιο αρκετά ευρύ. Και επίσης οι Ιαπωνέζοι συζητούν για εμπορική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Πώς επηρεάζουν οι συνομιλίες εμέν της ΔΕ. Μήπως πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς των δικών μας διαπραγματεύσεων τόσο να εξασφαλίσουμε την Ιαπωνία και μετά προχωρήσουμε προς την Κίνα. Υπάρχει έτσι κάποια πίεση. Και πώς το βλέπετε αυτό, πώς επηρεάζει. πώς επηρεάζει και τους Ιάπωνες τις συνομιλίες τους με άλλους. Μας είπατε τι προκλήσεις υπάρχουν στην Ιαπωνική αγορά. Εμείς μήπως θα πρέπει να κατεβάσουμε τον πύχη στον αφορά τις δικές μας προδιαγραφές για να μπορέσουμε να διεισδύσουμε στην Ιαπωνική αγορά. και τέλο πάντων κρατήσουμε ζεστό το ιαπωνικό ενδιαφέρον για μια συμφωνία μαζί μα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Όχι, όχι, δεν θέλω να σας ζωρίσω. Απλώς θέλω να με ενημερώσετε. Πώς βλέπετε το timing, το, το, το χρονισμό του αυτών των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, υπάρχουν πιθανότητες σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μετά τις διαπραγματεύσεις. Αυτό απλώς και μόνο. short Δύο σύντομες ερωτήσεις έχω. Γιατί προβληματίζεται τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την προτιμησιακή ρύθμιση αφού ήδη υπάρχει συμφωνία και για αυτά τα εμπορεύματα που θέλει να βγάλει από τον κατάλογο των ε, καλυπτωμένων προϊόντων, τον delisting. Όμως αυτό θα μας αποξενώσει την Ιαπωνία. Τι έχουν κάνει κάποια προσπάθεια την πρώτη χρονιά των διαπραγματεύσεων γιατί για το NTP ήδη συμφώνησαν. Μήπως θα ήταν καλύτερα να λάβουμε υπόψη την καλή πίστη των Ιαπωνέζων και να έχουμε κάποιο είδους συνεργασία μεταξύ των εταιριών Ιαπωνικών και δικών μας. Ήδη αυτό έχει αποδειχθεί ότι δουλεύει. Ε, αναφέρομαι στο συνδρομικό πακέτο. Ευχαριστώ. Τώρα έχω ακόμα έξι εγγεγραμμένους και κλείνω τον κατάλογο. Κύριος Προύστο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, το υπόθηκε και νωρίτερα, και αποφασίζει να διαπραγματευτεί ένα ε, σύνολο προτάσεων για τους σιδηροδρόμους, όπως πήγε ο κύριος Βαλένσα. Ρωτώ λοιπόν, τι είδους εντολή έχετε. Γιατί μόνος του ο Επίτροπος Ντεγκιούχτ ασχολείται με ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει γενικά τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω για τον delisting των τριών αυτών ε, φορέων των στερεοδρομικών επιχειρήσεων της Ιαπωνίας που ήταν δημόσιες επιχειρήσεις με συμμετοχή του Ιαπωνικού κράτους στο παρελθόν, τώρα είναι πλήρως θετικοποιημένες. Δέχεστε ωστόσο στους τρεις αυτούς ιδιώτες που ε, διακατέχουν το 60% της αγοράς να επαφεθούν τα ενία της δημόσιας επικοινωνίας, ενημέρωσης, ακόμα και των ξένων φορέων που θέλουν να μπουν στην αγορά. Το πιστεύετε και νομίζω ότι το παρελθόν είναι σαφέστατο. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα επιτρέψουν αυτοί οι Άπωνες ε, να συμμετάσχουν στην Ιαπωνική αγορά ξένοι και διευρωπαίοι. Ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε τόσο αφελείς. Επίσης μιλάτε για πλεονεκτήματα για την Ευρώπη. Σε λίγες όμως γραμμές. Το 90% αυτού του υπομνήματος αναφέρεται σε ε, λύσεις οι οποίες εξαρτώνται από την καλή βούληση και μόνο της Ιαπωνίας. Εάν θελήσει δηλαδή θα αφήσει πρόσβαση σε αγορές. Εσείς έχετε βάσιμους λόγους να έχετε αυτή την πεποίθηση για τις, καλές, για τις καλές προθέσεις. Μπορεί η Ιαπωνία να βρίσκεται μακριά. Αλλά επιτρέψτε μου για το θέμα αυτό να πω ότι η, Ελληνική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται πολύ πιο μακριά από την πραγματικότητα. Και τι νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε ότι εξασφαλίζουμε εάν αφήσουμε αυτούς τους τρεις παράγοντες επιχειρήσεις οι ιαπωνικές να ρυθμίσουν την αγορά χωρίς την παραμικρή εγγύηση. Οι Ευρωπαίοι δεν φαίνεται να έχουν συμμετάσχει στο πακέτο που προτείνεται. Τι ερωτήματα λοιπόν συγκεκριμένα έχετε διατυπώσει στο πλαίσιο της διαβούλευσης και αυτά είναι σύμφωνα με τόσα έχετε πραγματευτεί. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και με χαρά ακούω την ε, ενημέρωση για το τελευταίο αυτό στα διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι έχει σημασία να ασχοληθούμε με πολλά θέματα, όχι μόνο με το TTIP και βέβαια να μην εξαρτηθούν τα πάντα από μία και μόνο συμφωνία. Η Ιαπωνία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων, δεν πρέπει να είμαστε μόνο από τους Αμερικανούς. Αναφερθήκατε σε προθεσμίες και την προοπτική για το 2015. Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η εξέλιξη, το δεχόμενο δηλαδή να μην τηρηθεί το 2015 ως προθεσμία κατάληξης των διαπραγματεύσεων και τι είδους αλλαγές μπορεί να εμφανιστούν στον πολιτικό χάρτη της Ιαπωνίας μετά τις εκλογές του 2016. Επίσης τι ευκαιρίες αλλά και κινδύνους βλέπετε για τη γεωργία της, ε, ε, της Ευρώπης από αυτή τη συμφωνία. Κυρία Ρέντινγκ, θα ήθελα καταρχάς να πω ότι συμφωνώ απολύτως με την ερώτηση του κύριου Προύστου και θέλω να επισημάνω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά όχι μόνο το τι θα συμπεριληφθεί στο κείμενο αλλά και πώς θα υλοποιείται το κείμενο όχι μόνο δηλαδή υποσχέσεις αλλά και πραγματικότητα. Δεύτερη ερώτηση στα αγγλικά. Πολλά πράγματα διαπραγματευόμεθα. Η TTIP βεβαίω είναι ένα κομμάτι. Οι Ηνωμένε Πολιτείε όμω διαπραγματεύονται και μια ε, διειρηνική, δηλαδή πέραν του ειρηνικού, συμφωνία. Ε, υπάρχει κάποια συνέπεια και συνοχή σε όλες αυτές τις ε, εξελίξεις και τι είδους συντονισμός υπάρχει μεταξύ των διαπραγματευτικών μας ομάδων. Μπορεί να υπάρξει ένα σχήμα ρυθμιστικό τριμερές. Και στο θέμα των υπηρεσιών, τι είδους συντονισμός υπάρχει στις ε, συνομιλίες με την Ιαπωνία. Ευχαριστώ η Μαρίν Λεπέν. Η Ιαπωνία είναι μια χώρα της οποίας ε, συρρυκνούνται η οικονομία και θα συνεχίσει να συρρυκνώνεται και στο μέλλον και θα έχει πολύ χαμηλή ανάπτυξη αν το δούμε πολύ μακροπρόθεσμα. Ερωτώ λοιπόν αν είναι προς το συμφέρον μας η υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας. Η Ιαπωνία δεν κινδυνεύει να αρχίσει να εξάγει από εμά την ύφεση και τον αποπληθωρισμό. Εξάλλου είναι μια χώρα η οποία δύσκολα αποδέχεται ε, προϊόντα του, της Αλοδαπής ε, λόγω των πολύ ισχυρών πολιτικών ε, οικογενειακών της παραδόσεων όπως έχει άλλωστε καταδειχθεί και σε διάφορα βιβλία. Ε, πολλές φορές έχουν ειδικέ διατάξεις για την προστασία της ιαπωνικής αγοράς από ξένα προϊόντα και διερωτώ με αν είναι χρήσιμο να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε, να τους πιέσουμε να ανοίξουν αγορές μα τους δεδομένου ότι έχουν τόσο μεγάλη παραδοσιακή ε, νοοτροπία κλεισίματος και μήπως αυτό τελικά μας αποβεί ε, αποβεί βάρος μας. Τι άλλο μπορούμε να δούμε σε σχέση με το άνοιγμα της αγοράς της Ιαπωνίας και προς τους γείτονες. Μήπως ε, με, το, με την προσπάθεια για ένα ταυτόχρονο άνοιγμα όλων των μεγάλων οικονομιών διαπιστώνουμε τελικά ότι καμία χώρα δεν είναι διατεθειμένη να ανοίξει προς τους πάντες την αγορά της. Το θέμα δε των, της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ένα μελανό στίγμα σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις. Το 95% της, αυτοκίνητο, της αγοράς αυτοκινήτου της Ιαπωνίας το διακατέχουν οι άπονες παραγωγοί. Είναι οι πολύ συγκεκριμένες οι διατάξεις. Το 40% των πολλούμενων οχημάτων είναι τα μίνι οχήματα τα οποία δεν κατασκευάζουν οι Ευρωπαίοι. Είναι αδύνατον σχεδόν να μπει κανείς στην ευρωπαϊκή αγορά ή στην ιαπωνική αγορά. Οι όροι της βαθμονόμησης και της ε, ε, αντιστοιχεία των ισοτιμιών είναι πολύ διαφορετική ενώ η ιαπωνική αγορά είναι πολύ κλειστή, η ευρωπαϊκή είναι πολύ διαφανής και ανοιχτή και νομίζω ότι το να προσπαθήσουν να μπουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες μας στο, στην ιαπωνική αγορά μπορεί να αποβεί μπούμεραγκ αυτές και πολύ δυσμενές. Έτσι λοιπόν βλέπω ότι αυτές οι συμφωνίες για μια ε, για ένα απόλυτο άνοιγμα των εμπορικών ε, σχέσεων με την Ιαπωνία. Τεράστιο και βαρύτατο σφάλμα, αλλά δυστυχώ είναι φιλελεύθερη νοοτροπία. Σα το επιβάλλει. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, Ουρίγκα. Ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για όσα μας είπε, που ήρθε εδώ να μας εξηγήσει τα των διαπραγματεύσεων. Έχω κάποια θέματα που θέλω να σας θέσω πρώτα πρώτα. Έχουμε δει ότι η Ιαπωνία έχει αλλάξει ρότα στην εμπορική πολιτική. Όμως αυτές οι αλλαγές δεν είναι αυτές που θα θέλαμε κυρίως σε σχέση και με την ισοτιμία των νομισμάτων μας και βεβαίως είναι και θέμα ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας των Ιαπώνων δεν ξέρω τι μπορούμε να βάλουμε σαν ρήτρα στην συμφωνία. Αλλά βλέπουμε ότι το ζήτημα της ε, ζήτησης και προσφοράς των μικρών αυτοκινήτων είναι ένα πρόβλημα για την δίσδυση μας στην Ιαπωνική αγορά. Άρα όλα είναι και πιο σημαντικό το πώς θα έρθουν αυτοί οι σχετικοί φραγμοί. με τους μη δεσμολογικούς φραγμούς θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει γιατί οι βιομηχανίες αυτοκινήτων στην Ισπανία έρχονται σε επαφή μαζί μας και μας λένε το πρόβλημά τους. Θα πρέπει δηλαδή κάπως να προχωρήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση σχετικά με αυτό. Τώρα κάτι άλλο. Η κυρία Μάστρον όταν ήρθε για την ακρόαση που την αφορούσε ανέφερε το ότι μπορούμε να έχουμε κάποιες ρήτρες διαφύλαξης στην εμπορική συμφωνία. Για πέστε μας, γίνεται κάτι τέτοιο, να έχουμε δηλαδή ρήτρα διμερή διαφύλαξης στην συμφωνία με την Ιαπωνία και να έχουμε κάποια ίσως ε, μεταβατική περίοδο και τελικά κάποια στιγμή να γίνει ενεργοποίηση των ρητρών. Τι Όχι, τσίχου, τσίχου λέγομαι πρόεδρε. Eh, eh, πρόεδρε, θα πρέπει, νομίζω, να συγχαρούμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Γιατί μας έδωσε μια απεικόνηση πλήρη του τοπίου των διαπραγματεύσεων και θα πρέπει βέβαια να δούμε επί τη βάση των στοιχείων που μας είπε εάν ισχύουν όλα αυτά. Ε, λέμε ότι έχουμε αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρώπη 0,6 σε 0,8% και λέμε ότι θα έχουμε κάποιες εξαγωγές ε, προς την Ιαπωνία που θα είναι το 32% αυτού του ΑΕΠ και θα πρέπει επομένως να κάτσουμε και να δούμε ε, το πόσο, τι αντίκτυπο θα γι' αυτό αφού μιλάμε για το 4.000 και θέσεις εργασίας. Συγγνώμη, ναι, 3.200 θέσει εργασία θα δημιουργηθούν, οπότε θα πρέπει να κάτσουμε και να σταθμίσουμε τι, θα, επιπτώσεις θα υπάρχουν τελικά. Να σταθμίσουμε καλά τον αντίκτυπο της συμφωνίας. Νομίζω ότι προχωρά προσεκτικά η Επιτροπή και θα πρέπει να κάνουμε μια προκαταρκτική ε, μελέτη επιπτώσεων για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και στον αγροτικό τομέα. Σε 10 λεπτά θα πρέπει να μας απαντήσετε κύριε εκπρόσωπο της Επιτροπής. Είστε όλο και πιο φιδωλός με εμένα, Πρόεδρε. Ας ξεκινήσουμε το αυτοκίνητο. Που είναι ένα σοβαρό αυτοκίνητο από ό,τι φαίνεται. Επιτρέψτε μου να σα υπενθυμίσω ότι τα άνω των δύο τρίτων των Ιαπωνικών αυτοκινήτων που στην Ευρώπη είναι κατασκευασμένα στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να σα υπενθυμίσω ότι τώρα εξάγουμε πιο πολλά αυτοκίνητα προ την Ιαπωνία από όσα εξάγει η Ιαπωνία προ την Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να σα υπενθυμίσω ότι το πρωταρχικό πρόβλημα τη Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία έγκυται στην εσωτερική αγορά. Και επιτρέψτε μου επίση να μην ε, δεχθώ την ε, απόδοση στην Ιαπωνία όλων ε, των ε, προβλημάτων και των δεινών που γνωρίζει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Από την άλλη βεβαίως μπορεί αυτή η σχέση στις πωλήσει, το άνοιγμα των πωλήσεων μπορεί να φέρει σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο και με ιδιαίτερη προσοχή μελετάει τα ζητήματα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως άλλωστε ορίζεται και σαν την του Συμβουλίου για την διαπραγμάτευση για τις ανησυχίες του κυρίου Τσίκου. Αυτά τα βλέπουμε ήδη στην προκαταρκτική μας αξιολόγηση συνεπειών. Όπως έλεγα είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την υποβολή της προτάσεως για τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διαπραγματεύσεις προβαίνει στην αξιολόγηση των συνεπειών όπως κάνουμε εδώ και χρόνια για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ήταν όμως ένα θέμα περίπλοκο ε, διότι δεν είχαμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο εγχείρημα, αλλά μόνο με μία προβόλη, με μία υπόθεση για το τι περίπου θα περιελάμβανε η τελική συμφωνία. Πάντως, τα στοιχεία είναι αυτά τα οποία σας έχουμε υποβάλει. Θα ήθελα επίσης να, υπογρα... να υπογραμμίσω ότι οι συνθήκες αυτές ε, σημαίνουν ταυτόχρονα ότι με μια πολύ περιορισμένη συμφωνία δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε 150.000 θέσεις εργασίας και ιδιαίτερως και στην αυτοκινητοβιομηχανία αν δεν έχουμε δηλαδή πιο ευρύ πεδίο διαπραγματεύσεων άρα θα πρέπει αντίστοιχα να προσαρμοστούν τα στοιχεία αλλά τα στοιχεία που έχουμε υποβάλει εμείς είναι αξιόπιστα με βάση τις υποθέσεις μας ε, σαν υπόθεση εργασίας. Ε, το κύριο μέλημα νομίζω και το συμφέρον της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης να πολύ περισσότερα αυτοκίνητα και κυρίως περισσότερους τύπους αυτοκινήτων είναι αυτό που έχει να κάνει με την ομολογοποίηση. Όχι γιατί έχουν ριζικά διαφορετικές προδιαγραφές και πρότυπα οι Άπωνες, άλλωστε είναι ενεργό μέλος της Επιτροπής η ΕΝΙΣΗ και συμμετέχουν σε όλα τους κανόνες περιτυποποίησης και σε όλες τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις για τα αυτοκίνητα. Η Ιαπωνία υλοποιεί, εφαρμόζει τα πρότυπα αυτά κατά τρόπο λιγότερο τακτικό από ότι η ευρωπαϊκή πλευρά και μερικές φορές όταν το πράττει αυτό συμπεριλαμβάνει και προποθέσεις που δεν προβλέπονταν. Εκείνο είναι το πρόβλημά μας. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και εμείς πρότυπα αυτοκινητοβιομηχανίας και γι' αυτό δεν έχουν καμία δυσκολία οι Άπωνες να ε, πουλούν στην Ευρώπη και γιατί δεν χρειάζεται εμείς να προσαρμόζουμε τα πρότυπα. Μας έχουμε κοινά πρότυπα δηλαδή. Αυτό που θέλουμε πάντως να επιβάλλουμε είναι μια πλήρης και αυστηρή τήρηση των διεθνών προτύπων και ενισχυμένη συνεργασία κατά τη διατύπωση των νέων προτύπων όταν εξελίσσονται τα οχήματα. Ε, υπ' αυτή την έννοια και από τη δική μας την προοπτική υπάρχει και η ε, έννοια της ευρύτερης συνεργασίας με άλλους ε, αυτοκινητοπαραγωγούς ανά τον κόσμο Ιδιαίτερο των ΗΠΑ. Ένα εγχείρημα που δεν είναι ευχερέ γιατί οι Αμερικανοί έχουν διαφορετική αντίληψη ω προ τα διεθνή πρότυπα για τα αυτοκίνητα από αυτή που έχουμε εμεί οι Άπωνε. άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε θαύματα βραχυπρόθεσμα, πάντως παραμένει ανοιχτή η επιλογή. Επίση αληθεύει ότι υπάρχουν και άλλα εμπόδια σε σχέση με τι ε, εμπορικές συναλλαγέ με την Ιαπωνία, η διανομή έχει συζητηθεί. Οι, οι έχουν, κάνει, έχουν προβεί σε μονομερείς παραχωρήσεις το θέμα της διανομής. Εμείς θα έχουμε σε εκ τούτου καλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη δικτύου διανομής στην Ιαπωνία από αυτή την έννοια. Και είναι λυπηρό το ότι αυτή η ευκαιρία έχει αξιοποιηθεί από ορισμένου εισαγωγείς ευρωπαϊκών αυτοκινήτων αλλά η αυτοκινητοβιομηχανία ευρωπαϊκή έχει ζητήσει την αξιοποίηση των νέων αυτών κανόνων για να μπορέσει να ιδρύσει ένα, ένα σύστημα δίκτυο διανομής στην Ιαπωνική αγορά. Όπως σας είπα είναι αυτά τα ποσοστά για την συμμετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας ε, και τα ωφέλη τα φορολογικά που προβλέπονται όταν πρόκειται για μικρά αυτοκίνητα. Πληθυσμό στην, Ήπεθρο, κοινωνικά κίνητρα και ειδική μεταχείριση εκτίου του για κάποιε κατηγορίε αυτοκινήτων. Αυτό που προσπαθούμε να πείσουμε του Ιάπωνε είναι ότι μπορούν οι ίδιοι στόχοι να εκπληρωθούν και με διαφορετικό τρόπο και ότι μπορεί να υπάρχουν συμπληρωματικοί σημαντικοί στόχοι όπω η καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση των αυτοκινήτων οι οποίε ε, ξεφεύγουν, δεν εξυπηρετούνται απαραίτητα από τα φυσικά ε, οι μηχανικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα το δεχθούν. Ε, ίσως να μπορέσουμε να το βάλουμε σε μια συμφωνία, αλλά δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε σε μια εμπορική συμφωνία την φορολογική βάση και τα ποσοστά, του συντολεστέ, του φορολογικούς. Δεν ήταν καν η εντολή μας, ούτε νομίζω ότι θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε αποστολή και εντολή διαπραγμάτευση σε θέματα θεμάτων φορολογικών μέσα σε μια εμπορική συμφωνία. Αλλά ίσως αυτό να πείσει του Ιάπωνες ότι θα μπορούσαν να κάνουν μια προσαρμογή ω προ τη φορολογική τους βάση και του συντελεστέ για να προωθήσουν μια συμφωνία με τους Ευρωπαίου. Δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι ικανοποιητικά τα πάντα ως προς την ε, υπόθεση αυτή, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα βελτιώσουμε. Στις δημόσιες προμήθειες που είναι επίσης άλλο αμφιλεγόμενο ζήτημα. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι μια ιδιωτική εταιρεία ή ουδήποτε τύπου δεν υπάγεται στους ε, κανόνες περί δημόσιων προμηθειών. Οι εν λόγω τρεις ιαπωνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ε, υπαχθεί σε οποιαδήποτε εθνική ή διεθνή υποχρέωση περί δημοσίων προμηθειών η διάταξη εδώ και χρόνια. Εμείς, και επειδή μας κατηγορούν οι Άπωνες ότι δεν έχουμε ισότιμη αντιμετώπιση, εμείς καταγράφουμε τις επιχειρήσεις αυτές ε, αποκλείοντάς τις από τον κατάλογο του GPA, των γενικευμένων προτιμήσεων, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι ικανοποιητικό ο τρόπος με τον οποίο τις χειρίζονται οι Ιάπωνες. Δεν βλέπουμε δηλαδή τι ισχύει, πώς μπορεί να ισχύσει, πώς μπορούν οι προϋποθέσεις ασφαλείας τις οποίες ζητούν οι Ιάπωνες να ισχύσουν για τους δικούς μας παραγωγούς, για τις δικές μας επιχειρήσεις, αλλά πάντως η επίπτωση ήταν μηδενική, μηδενικός αντίκτυπος. Τίποτε, ουδέν δεν μπορούσε να έχει ε, αντίκτυπο πρακτικό στο εμπόριο αυτή η αντιμετώπιση παρά μόνο πολιτικό γιατί βλέπει η Ιαπωνία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τη μεταχειρίζεται κατά τρόπο διαφορετικό από ότι οδήποτε άλλη χώρα ανοίξει το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων. Και αυτό το πράξαμε διότι θεωρούμε ότι δεν έχουμε ούτε αυτή ισότιμη αντιμετώπιση στο ίδιο θέμα. Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων ε, οδηγεί σε ένα πακέτο το οποίο μας κάνει να βγάλουμε αυτήν την άνηση μεταχείριση, επειδή έφυγε και από την άλλη πλευρά η άνηση μεταχείριση. Οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή θεωρούν ότι έχουμε φτάσει στο στόχο μα, γιατί ο στόχο μα δεν ήταν να αυξήσουμε την πρόσβασή μα ε, στην Ιαπωνική αγορά δημοσίων προμηθειών. Αυτός ο στόχος είναι ουσιώδης, είναι θεμελιώδης, ο των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να επιτευχθεί ασφαλώς και δεν νομίζω ότι μπορεί να υποβληθεί από πλευρά της Επιτροπής ε, σχέδιο συμφωνίας με την Ιαπωνία χωρίς να περιλαμβάνει αυτό σχέδιο για ένα εύλογο βέβαια άνοιγμα των Ιαπωνικών αγορών δημοσίων προμηθειών. Αλλά το θέμα αυτό δεν είναι μόνο τη Shinkansen, δεν είναι των τριών αυτών επιχειρήσεων, είναι, το, ε, είναι η, η συμβατική σιδηρόδρομη, η ελαφρύ σιδηρόδρομη, ε, το τραμ και τα άλλα μέσα σταθερής τροχιάς. Όλα αυτά θα ωφεληθούν από υποχρεωτικούς διαφανείς κανόνες και όλα αυτά θα, έχουν, θα πρέπει να επαχθούν στην, στις διατάξεις για την πρόσβαση στην αγορά. Από εκεί άλλωστε θα υπάρξει και το κύριο κέρδος. Δεν νομίζω ότι θα πωληθούν πολλά προϊόντα της Shinkansen στην Ευρώπη, όπως θα δούμε και πολλά της TGV να πολλούνται στην Ιαπωνία, αλλά αυτό είναι κλάσμα μόνο της ε, παραγωγής ε, της βιομηχανίας σιδηροδρόμων της Ευρώπης. Και εμεί κινούμαστε με στόχο να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα όλη τη βιομηχανία σιδηροδρόμων. Έχουμε διαβουλευθεί με, την, ε, με τον κλάδο, ο οποίο μα έχει πει ότι ο μακροσκελή κατάλογο που έχουν υποβάλει οι Ιάπωνε συνεπάγεται προβλήματα ω προ προς τις συνθήκες ασφαλείας. Θα πρέπει να δούμε εμείς αν θέλουμε, εάν μας χρειάζεται το κεφάλαιο που αφορά την ε, ασφάλεια. Ε, ευσταθεί αυτό που υπόθηκε ότι στηρίζεται στην ε, καλή πίστη της Ιαπωνίας συμφωνία, όπως όμως στηρίζεται και στην καλή πίστη των Ευρωπαίων, χωρίς καλή πίστη καμία συμφωνία δεν μπορεί να ισχύσει, μόνο από την Χάνον. Και για να ξαναγυρίσω στι ε, προμήθειε, θα ήθελα να πω ότι αυτή η συμφωνία για του σιδηροδρόμου επισκιάζει το γεγονό ότι έχουμε τεράστια συμφέροντα για άνοιγμα των δημοσίων προμηθειών στην Ιαπωνία σε τόσου άλλου τομεί που δεν μπορέσαμε ακόμα να ανοίξουμε τη συζήτηση με του Ιάπωνε λόγω ακριβώ των προβλημάτων και των στόχων για του σιδηροδρόμου. Και γι' αυτό ακριβώ περιμένω τη μέρα που θα μπορέσω να διαπραγματευτώ με του Ιάπωνε το μεγαλύτερο κομμάτι των οικονομικών μα συμφορών χωρί να χρειάζεται να κολλάω σε έναν υποτομέα ενό τομέα που μπορεί να είναι και τα συμφέροντα μια μόνο και μεμονωμένη επιχείρηση. Και Κατά τα άλλα, με πολύ μεγάλη χαρά ε, θα δώσω επιμέρους απαντήσεις σε διμερείς επαφές, εάν θέλουν οι ίδιοι βουλευτές ή οι, βουλευτές, οι βοηθοί τους. Δεν θα μπορούσα δυστυχώς να μπω σε όλες τις ε, λεπτομέρειες. Για το χρονοδιάγραμμα, ε, το 2015 είναι λογικό χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, πιστεύω ότι μπορούμε, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα το πράξουμε, θα τα καταφέρουμε. συνέπεια, συνέπεια του να μην τηρηθεί αυτή προθεσμία. Είναι άγνωστον, δεν μπορούμε να την αξιολογήσουμε αυτή τη στιγμή και δεν έχω καμιά όρεξη να προβλέψω την έκβαση των Ιαπωνικών εκλογών του 2016. Εάν ο Πρωθυπουργό Άμπε κερδίζει τι εκλογέ, βεβαίω θα έχουμε τον ίδιο εταίρο. Ο διάδοχό του όμω ενδεχομένω να έχει διαφορετικέ απόψει ή και τι ίδιε. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι είναι πολύ σημαντικό ο, για το πρόγραμμα εσωτερικών μεταρρυθμίσεων του Πρωθυπουργού Άμπε να ολοκληρωθούν αυτές τις πραγματεύσεις με τη σύναψη της σύμβασης και αυτή η σύναψη της σύμβασης δεν μπορεί να γίνει κατά τρόπο που δεν ευθυγραμμίζεται με τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Έτσι άλλωστε λειτουργεί και η εσωτερική αγορά, έτσι και μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε στη σύναψη αυτής της σύμβασης, επομένως της συμφωνίας. Επομένως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Λοιπές διαπραγματεύσεις. Σαφής ε, παρεμβολή της ε, ITTP υπάρχει ασφαλώς από πλευρά των Αμερικανών που θέλουν να επιβάλλουν, ε, να παρισφρήσουν και να επιβάλλουν τα δικά τους συμφέροντα. Έχουν διαφορετική θεώρηση σε πολλά πράγματα. Περιορισμένος συντονισμός μεταξύ διαπραγματευτών διαφόρων κρατών. Με τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις δεν έχουμε πολύ περιθώριο παρά μόνο για την εγωιστική προσέγγιση. Οι παρεμβολές αυτές νομίζω ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν βλέπουμε ιδιαίτερη παρεμβολή και ε, επίδραση των διαπραγματεύσεων αυτών ε, της Ιαπωνίας σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα και Τούμπαλιν. Πρόεδρε, ξέρω ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, ξέρω ότι έχω δυσαρεστήσει αρκετούς από εσά, όπως έλεγα. Μπορώ να δώσω τις απαντήσεις διμερός σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι δεν καλύφθηκε σε αυτό το στάδιο. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Είμαι σίγουρο ότι θα έχουμε και ευκαιρία να τα πούμε μαζί σα όσον αφορά τι ε, Ιαπωνο-Ευρωπαϊκές σχέσεις. Τώρα δύο λόγια από τον εισηγητή μα. Ναι, Πρόεδρε, εντάχει, να ευχαριστήσω τον κύριο Πετρουτσάνη για ε, όσα μα ε, εξήγησε, για όσα μα απάντησε. Όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ διαφορετική προβληματική. Και όντως έχουμε τώρα μια μοναδική ευκαιρία στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου. Πάντως με ευχαρίστηση άκουσα ότι θα γίνουν ε, επιπλέον πρόσθετες διαπραγματεύσεις κατόπιν της πρόοδο που ήδη σημειώθηκε. Βεβαίω και θα επανέλθουμε στο θέμα. Συγκεκριμένα μετά τον 7ο γύρο διαπραγματεύσεων. Και θα υπάρχει επίση και διακοινοβουλευτική συνάντηση κάποια στιγμή φέτο. Συναδελφοί, στις 12 θα αρχίσουν ε, ε, οι συντονιστέ στη ζήτησή του. Τώρα έχουμε ένα πραγματικά σημαντικό θέμα, το θέμα της Ουκρανίας. Πρόκειται για την προτιμησιακή συμφωνία εμπορικών με την Ουκρανία στα γερμανικά. Σε σχέση λοιπόν με την Ουκρανία και τη Συμφωνία Σύνδεσης Εταιρικής Σχέσης έχουμε μία συζήτηση διεξαγάγει εισαγωγικά γιατί ετέθη το ζήτημα της αναβολής της εφαρμογής Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ουκρανία με συναφέ ζήτημα την απέτηση για την Επιτροπή να παραταθούν οι γενικευμένες προτιμήσεις με την Ουκρανία που θα έπρεπε να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου εφέτος. Η δυνατότητα αυτή είναι πρωτοφανής, δεν την είχαμε στο παρελθόν. και ως εκ τούτου είχαμε και δύο πρόσθετες απαιτήσει. Αφενός μεν σε άλλα σημαντικά θέματα γενικευμένων εμπορικών, προτιμ... Ε, εμπορικών προτιμήσεων να προχωρούμε με βάση τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στην αναγνώριση των προτιμήσεων, των ανθρωπινών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων ε, ή των αρχών του κράτους δικαίου όπως άλλωστε προβλέπεται και ρητά στην Συμφωνία Σύνδεσης. Προϋποθέσεις λοιπόν θεμελιώδεις, οι οποίες πληρούνται. Προϋπόθεση θεμελιώδης, η οποία ε, πληρείται πιστεύω. Έχει συμπεριληφθεί στις ε, εμπορικές προτιμήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε στην αρχή του χρόνου επισημάνει. Και επίσης κάτι άλλο είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε τι, ε, τι αντίκτυπο έχουν αυτές ή μπορεί να έχουν αυτές οι προτιμήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα έπρεπε να προβεί σε μια αξιολόγηση των οικονομικών συνεπειών των εμπορικών προτιμήσεων ώστε και εμείς να γνωρίζουμε για τη δική μας οικονομία τι είδους συνέπειες μπορεί να επιφέρουν αυτές. Με βάση λοιπόν αυτά. Θέσαμε, έστω και τελευταία στιγμή, το θέμα αυτό στην εμμυρίσια διάταξη και προβλέψαμε τη δυνατότητα να γίνει μια απλουστευμένη διαδικασία ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να αντιδρούμε εγκαίρως. Ο πρέσβης της Ουκρανίας μου απέστειλε μια επιστολή όπου υπογραμμίζει τη σημασία μιας ε, ταχείας και πρόσκοπτης διαδικασίας και ταυτόχρονα δηλώνει ότι σκοπεύει να τηρήσει τις δεσμεύσεις ανά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον, έχω λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον προεδρεύοντα καλύτερα, τον Ιταλό, όπου με ενημερώνει για την, πρόστα... για την συζήτηση στις 26 Σεπτεμβρίου της προτάσεως να μην... Ε, όπου κανένα μέλος εκ των 28 κρατών μελών δεν αντετέθη στην πρόταση. Και ως εκ τούτου, οι δύο ισιώδεις προϋποθέσεις που είχαμε διατυπώσει διαπιστώνουμε ότι έχουν εκπληρωθεί. Αυτό ισχύει και για την Ουκρανία, αλλά και για τα 28 κράτη-μέλη, φαίνεται ότι συμφωνούν σε αυτό, γιατί βλέπουμε μια ομόφωνη θέση υπέρ της προτάσεως. Στο βαθμό αυτό, εφόσον συμφωνείτε, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια απλουστευμένη διαδικασία Μία έκθεση δηλαδή χωρίς τροπολογίες στην Ολομέλεια. Είναι μια επιλογή την οποία θα ε, ψηφίσουμε, θα εγκρίνουμε με την ψήφο μας στο τέλος της συζήτησης. Διαδικαστικό, Πρόεδρε. Με ποιο άρθρο του, ε, του κανονισμού, ποιο άρθρο του κανονισμού επικαλείστε. Ναι, για την ψηφοφορία, Πρόεδρε. Σε 20 λεπτά περίπου. Προβλέπετε την ψηφοφορία. Ίσως δεν κατάλαβα. Ο πρόεδρος. Ε, ορίσαμε την ημερήσια διάταξη στην αρχή της συνεδρίασης. Και είπαμε για το σημείο 12, ανταλλαγή απόψεων και πιθανή ψηφοφορία. Πιθανή όμως είναι, σημαίνει κάτι άλλο. Εγώ θέλω να καταλάβω τι συμβαίνει. Δεν θα δεν σας ε, κατακρίνω. Δηλαδή μου λέτε ότι θα γίνει ψηφοφορία. Κάπου στις 12 παρα 5 αυτό μου λέτε πρόεδρε. Το όντι λέει ο πρόεδρος. Μου το λέτε και στα αγγλικά. Ε, και, και γερμανικά μιλάτε έτσι. Μιλάω μάλλον. Μιλάτε και εσείς. Μπορείτε να πείτε «για», μπορείτε να πείτε και «nein», «aber», θα ήθελα να καταλάβω. Ναι, βεβαίως. Εάν συμφωνήσουμε σε μια απλουστευμένη διαδικασία, θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε ψηφοφορία. Ε, διαδικαστικό, λοιπόν, θα, θα καλέσω, Πρόεδρε, να αναβληθεί η ψηφοφορία. Πρέπει να συλλέξω τα μέλη της ομάδας μου. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Δεν έχουμε ενημερωθεί εγκαίρως. Να προτείνω να είναι λίγο πιο οργανωμένη η συζήτηση να κάνουμε. Πρώτα μια συζήτηση να δούμε πώς θα πάει και ίσως αυτό θα μας δείξει κατά πόσο χρειάζεται τελικά να γίνει ψηφοφορία ή όχι. Γιατί και εμείς θα χρειαστεί να συλλέξουμε τα μέλη της πολιτικής μας ομάδας τώρα τελευταία στιγμή αν τελικά φανεί ότι χρειάζεται ψηφοφορία και ίσως να μην χρειαστεί αυτό, ίσως να υπάρχει συνένεση. Τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτό, θα, θα επανέλθω όταν έρθει ο, ο χρόνος που να μιλήσω. Ακριβώς αυτό θα πράξουμε, δεν είναι υποχρεωτικό να... Και έχω και άλλο διαδικαστικό, Πρόεδρε. Ποια είναι η απαρτία που απαιτείται για, για να γίνει ψηφοφορία, τι λέει ο κανονισμός. Τι λέει ο κανονισμός, προϋποτίθεται ελάχιστος αριθμός, να αρχίσω να μετράω κι εγώ. 11 βουλευτές για την απαρτία και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Για την απόρριψη της προτάσεως τέσσερις ψήφοι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρώτο. Παρακαλώ εσείς. Ο κύριος Λαντσμπέρκης. Uh, indeed you mentioned that uh, we have an extraordinary situation uh, regarding... Η κατάσταση φυσικά είναι εξαιρετική, είναι ιδιαίτερη. Δεν είναι συνήθις, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά δεν είναι και πρώτη φορά. Έτσι. Το έχουμε συζητήσει και στο Στρασβούργο, όταν υπερψηφίσαμε τη συμφωνία. Η γενικότερη κατάσταση στην Ουκρανία θα έλεγα ότι είναι εξαιρετική. Ε, εξαίρεση μάλλον. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε λοιπόν που συμπεριλάβατε αυτό το θέμα στην ημερησία διάταξη γιατί αυτή τη στιγμή το, η, Ουκρανία παλεύει για την εδαφική τη ε, κυριαρχία γιατί έχει να αντιμετωπίσει τεράστια οικονομικά προβλήματα, χρειάζονται μεταρρυθμίσει Επίση, Η Ευρώπη έχει δεσμευτεί να βοηθήσει την Ουκρανία γιατί είναι μια χώρα με την οποία γειτονεύουμε και θέλουμε να του βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να αντισταθούν στις πιέσεις οι οποίε θα μπορούσαν να οδηγήσουν όχι μόνο στο να μην ε, προχωρήσει η συμφωνία, αλλά και να παγώσουν οποιασδήποτε μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει λοιπόν η πρόταση για 15 μήνες να παγώσει η εφαρμογή της συμφωνίας. Πολλοί από εμά μας έχει, έχει απογοτεύσει αυτό, ωστόσο. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους Ουκρανούς, ε, ε, επεκτείνοντας τη συμφωνία για, τις, για τους ATMs, να βοηθήσουμε παρά το γεγονό ότι υπάρχει δυνατότητα ε, εφαρμογή εκ των υστέρων, εάν δεν επεκταθεί η συμφωνία, ε, θα δημιουργηθεί πρόβλημα, πρόβλημα στις επιχειρήσεις. Η ουκρανική πλευρά ισχυρίζεται ότι οι ATM έχουν βοηθήσει τις εξαγωγές της Ουκρανίας Κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτή τη στιγμή για τους Ουκρανούς παραγωγούς να αυξήσουν τις εξαγωγές τους προς την ευρωπαϊκή αγορά. Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, η κατάσταση στην Ουκρανία, όπως γνωρίζετε, δεν είναι μια συνήθις κατάσταση. Μας δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που θα κάναμε από φυσιολογικές συνθήκες. Γι' αυτό θα πρότεινα στις 12 Οκτωβρίου, εάν όχι σήμερα, να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα και αμέσως μετά να υπάρξει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια έτσι ώστε να επεκταθεί η ισχύ στον ATM. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ποτέ δεν μου άρεσαν οι συντοβεμένες διαδικασίες. Όμως ε, πολύ σωστά λέει ο συνάδελφος, δεν πρόκειται περί ε, καταστάσεως που ισχύουν πράγματα κάτι εξαίρεση και δεν είναι θέμα τώρα να ε, δούμε τι θα γίνει με τις ε, με, με, με, την, με, το να γεφυρώσουμε το, το κενό μεταξύ των προτιμησιακών ρυθμίσεων και της συνολικής συμφωνίας θα πρέπει προσωρινά να βρούμε κάποια λύση και θα πρέπει να δράσουμε ταχαίως γιατί πρώτη ενδεκάτου εκπνέει η ισχύουσα συμφωνία το οποίο θα φέρει αφεβαιότητα στους συναλλασσομένους ξέρουμε τις πρόστριβες με τη Ρωσία και άρα θα πρέπει να δώσουμε εμείς ένα μήνυμα, να στείλουμε ένα μήνυμα να συνεχίσει να είναι ανοιχτή για μας η αγορά της Ουκρανίας και άρα θα πρέπει να εγκρίνουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα το συντομευμένο. Έχουμε και το άρθρο 2. Έχει τώρα μια ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι τόσο κατοχυρμένο όσο θέλαμε, αλλά τουλάχιστον υπάρχει καταρχήν αυτή η ρήτρα. Ο επόμενος. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιδείξει ευελιξία και το θεωρούμε πολύ θετικό και Νομίζω ότι το σύστημα γεννημένων προτιμήσεων είναι κάτι το οποίο δεν μας κοστίζει αλλά είναι πολύ σημαντικό για την Ουκρανία γιατί έχουμε κάποιους ε, βασικούς υπολογισμούς ε, των εξαγών και μιλάμε για 10-20% των εξαγών μας που θα ρυθμιστούν έτσι κάτι το οποίο τέτοιες ώρες είναι σημαντικό για την Ουκρανία. Επομένω τα πάντα μπορούμε να πούμε τώρα ότι είναι κατεξαίρεση ρυθμίσεις και νομίζω επίσης ότι είναι θετικό να μπορέσει να διασκεδάσει τις αμφιβολίες μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι αυτές οι λύσεις που θα δοθούν τώρα θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Εννοείται ότι υπάρχουν και πιέσεις από πλευράς Ρωσίας. Τώρα κάτι άλλο. Μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν θα επιτρέψει ή όχι δυσμενείς αναθεωρήσεις των συμφωνιών σύνδεσης γιατί ξέρουμε πόσο έχει πιέσει επ' αυτού η Ρωσία. Μαρική. Όντως η κατάσταση ε, είναι μια κατάσταση έκτακτη κατ' εξαίρεση ενισχύουσα. Είδατε τι έγινε από το Σεπτέμβριο που τα πρώτο είπαμε και τώρα έχουμε αυτή την σπάνια ευκαιρία. Και εγώ θα πρέπει να σας πω τους προβληματισμούς μου μας ενημερώνει η Κομισιόν την 12η ώρα για τις τριμερείς επαφές Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης μας λένε ότι οδήγησαν στην αναστολή ε, ε, των εμπορικών ρυθμίσεων της Συμφωνίας σύνδεση. Αυτό είναι τελεσμένο γεγονός, τέτοιου είδους τακτική, ότι δηλαδή τώρα η κατάσταση δεν επιδέχεται μεταβολή και όλα αυτά είναι δύσκολα να, να, τα, να κρίνουμε να, και να ψηφίσουμε γιατί δεν ξέρουμε ένα σωρό ε, λεπτομέρειες. Παρακαλώ, θέλω να γραφεί στα πρακτικά ότι πιστεύω ότι αυτό που έγινε είναι πάρα πολύ δυσάρεστο αλλά δεν θα πρέπει να επανελευθεί. Δεν θα πρέπει ε, σαν ένας νταΐς η Ρωσία να επιβάλλει τις ρυθμίσεις που θέλει. Δεν θα πρέπει αυτό να επανελευθεί. Και δεν είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μαθαίνει από τι εφημερίδε τη εξελίξη Αντί για του ε, συνήθει κανονικού διάβλου. Ελπίζω ότι αυτή η διευθύνουσα επιτροπή, η steering committee, πρόκειται κάτι να κάνει και εσείς να το ε, ρυθμίσετε και να δούμε ε, να μείνει στις δεσμεύσει υποψηφία επίτροπο. πάντω η κατάσταση σε σχέση με την Ουκρανία τώρα είναι πάρα πολύ λεπτή, δύσκολη. Δεν είναι δυνατόν μια τέτοια κατάσταση να ε, εμποδίζεται από διαδικαστικά. Νομίζω ότι η πιο σωστή αντιμετώπιση είναι να έχουμε απλουστευμένη διαδικασία. Επίσης, νομίζω η ομάδα μας θα συμφωνήσει με τις προτάσεις ούτως ώστε να μην εμποδίσουμε τους εμπορευόμενους και από τις δύο πλευρές. Να μην έχουν να αντιμετωπίσουν αχρίαστα εμπόδια και δυσκολίες. Πάντως, προσοχή να μην αποτελέσει ένα προηγούμενο αυτή η κατάσταση και αντιμετώπιση. Δεν θα πρέπει να ε, άγεται και φέρεται το κοινοβούλιο και να αναγκάζεται να δώσει το πράσινο φως μηχανιστικά σε κάποιες αποφάσεις που η ίδια η Κομισιόν εξαναγκάζεται και από άλλους να λάβει. Να τα συζητήσουμε με τη νέα Επίτροπο να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις ε, επιθυμητές διαδικασίες. Φοβάμαι ότι δεν είναι τελευταία φορά που το εμπόριο πολιτικοποιείται και ότι εμείς πρέπει να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Πρόεδρος. Ως πρόεδρος της Επιτροπής μας δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω τόσο με κύριε Σχάκη. Ο κύριος Σόλτς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Βεβαίω είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το έχουμε συζητήσει το πώς θα πρέπει να χειριστούμε τα ζητήματα και την προηγούμενη φορά όταν μονομερός ε, εγκρίθηκαν ε, από την Επιτροπή κατά τρόπο πλειοψηφικό αυτά τα μέτρα, είπα ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε με μεγάλη προσοχή τι είδους συνέπειες θα έχουν για τις ε, οικονομίες των δύο πλευρών. Και πριν τοποθετηθώ εδώ θα ήθελα η Επιτροπή να μας ενημερώσει τι γίνεται ως προς τη συμβατότητα των μέτρων αυτών με τους ε, κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, πρώτον. Δεύτερον, ποια είναι τα ακριβή οικονομικά στοιχεία για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την, σε περίπτωση ε, εγκρίσεως και θέση εφαρμογή από απολεσθέντες δασμούς. 600 εκατομμύρια το εξάμεινο βλέπω εδώ, 1,5 δις λιγότερα έσοδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε και να ξέρει και ο πολίτης τι τον περιμένει. Θέλουμε τα τελευταία λοιπόν στοιχεία και τα πιο επίκαιρα. Τρίτον. Και η κυρία Σάκ το έθιξε το ζήτημα των τριμερών επαφών. Ποια είναι η κατάσταση Γνωρίζουμε ότι γίνονται τριμέρεις επαφές μέχρι εκεί. Το γεγονός το γνωρίζουμε, αλλά στο περιθώριο, στους διαδρόμους και κλεισμένων των θυρών τι συζητείτε δεν ξέρουμε και θέλουμε για να είμαστε και υπεύθυνοι σε αποφάσεις που θα λάβουμε να ξέρουμε πώς έχει ε, προχωρήσει η υπόθεση αυτών των διαπραγματεύσεων, ποια είναι η στάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ε, τι κάνουμε εμείς και τι περιμένει βέβαια τον Ουκρανικό λαό, μια και επέρχεται και ο επίκειται και ο χειμώνα και τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς τι είδους συνέπειες θα δούνε από πλευράς της Ρωσικής, ε, των σχέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Επίσης ε, θεωρώ ότι η επιταχυμένη διαδικασία, απλουστευμένη διαδικασία αποτελεί ε, παρέκβαση από τις δημοκρατικές αρχές και δεν την υποστηρίζω. Πρέπει να έχουμε όσο δυνατόν πιο ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες για να αποφύγουμε την απώλεια εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μέχρι τώρα μόνο την έχουμε υποσκάψει. Ω εκ τούτου, θέλω να μα κοινοποιήσετε την επιστολή του Ουκρανού πρέσβη. Ευχαριστώ. Γιάννη του. Δεν συμφωνώ μαζί σου, Χέλμουτ, όσον αφορά το ζήτημα των επιτυχημένων διαδικασιών. Όταν υπάρχει μια εκτακτή κατάσταση, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γενικότερα ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, έχουν την ε, δυνατότητα να παρέμβουν σε μια χρονική συγκυρία, εκεί πρέπει να το κάνει γιατί αυτό απαιτούν από, εμά, από εμάς οι πολίτες. Έχουμε ασκήσει κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονό ότι δεν έχουμε την επαρκή πληροφόρηση για την απόφαση που έλαβε το Σεπτέμβριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να παρέχει τις πληροφορίες που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται, έχει ανάγκη για να λαμβάνει τα μέλη του αποφάσεις πλήρως ενήμεροι και όλες τις πληροφορίες τις οποίες ζητούμε. Γιατί ο στόχος φυσικά είναι να καταφέρουμε να προσαρμοστούμε σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη και δύσκολη πολιτική κατάσταση. Είναι σαφές ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και έλλειψη πληροφόρησης. Γνωρίζουμε ότι η απόφαση του Σεπτεμβρίου, αυτή η αναβολή, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την πίεση από τη Ρωσία. Το ερώτημα λοιπόν είναι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αφήσει και άλλο χώρο στη ρωσική πλευρά. Θα δείξει ε, με αυτόν τον τρόπο ότι είναι ευάλωτο. Εγώ δεν το πιστεύω. Αντιθέτω, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να δεχτούμε αυτή την επιτυχημένη διαδικασία, η οποία σίγουρα δεν είναι τέλεια, αλλά η πολιτική συγκυρία σήμερα μα υποχρεώνει να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι ο πολίτη θα το αντιληφθεί παρά το γεγονό ότι δεν είναι η ορθή, η ενδεδειγμένη, συνηθισμένη. Γιατί διαφορετικά τίθεται σε κίνδυνο η διαδικασία εκδημοκρατισμού τη ίδια τη Ουκρανία. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι κατέστησα νωρίτερα σαφέ ότι αντίκειμε σε αυτή τη διαδικασία του να κάνουμε βεβαιασμένε αυτέ τι κινήσει και μάλιστα τόσο πολύ που όπω είδατε, ακόμα και γερμανικά μπορώ να τα πω. Και στο συγγνώμη, ή κάπω να τα πω. Ζητώ τα συγγνώμη όμω για την προφορά. Ε, επί τη ουσία όμω. Η δική μα θέση ήταν πάντα ότι η κατάσταση στην Ουκρανία είναι πολύ λεπτή οι, ο, οι ε, που μετέφερ, μετέφεραν τον κύριο που χρησιμοποίησαν τη λέξη fragile, χαζίλα, εύθραυστη, φαντάζομαι από τα γαλλικά, είναι έως και εκρηκτική. Η κατάσταση στην Ουκρανία το έχουμε καταστήσει σαφές έναντι κάποιων ε, φιλοπόλεμων βουλευτών του ΕΛΚ, αλλά και σοσιαλιστών πρέπει να πω, και πάνω απ' όλα πρέπει να πω ότι με καταπλήσει το γεγονό ότι η Επιτροπή συμφωνεί μαζί μα. Ότι αυτή η συμφωνία έχει εκρηκτικό περιεχόμενο ή συνέπειε και προτιμάει να την αναβάλει. Τουλάχιστον για ένα διάστημα. Είναι λοιπόν αξιόλογο το ότι οι Άλντε για μια φορά φαίνεται να διαφωνούν με αυτά που κάνει η Επιτροπή. Και έτσι θεωρούμε ότι σε μια κατάσταση εύθραυστη, λεπτή ισορροπία το να εισάγεται μια εκρηκτική συμφωνία αποτελεί πολύ επικίνδυνο συνδυασμό. Πιστεύουμε ότι μπορεί να προσπαθήσετε να το παραχώσετε την τελευταία στιγμή στην ημερήσια διάταξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το παραγνωρίσουμε εμεί. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Η κυρία Λεπέν έχει το λόγο. Δύο λόγια. Πρώτα πρώτα όσον αφορά την τετρατονομή δικαιωμάτων. Δεν ξέρω ότι είναι για γέλια, των για κλάματα. Γιατί είδατε τι γίνεται στις ε, πύλες της ε, Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κάτι για το οποίο κανένας δεν μιλάει. Πρόκειται για μια ομερτά, ένα blackout στα ε, μέσα ενημέρωσης της ε, Ευρώπης και της Γαλλίας βέβαια. Και αφού μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, να μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν πολιτισμοί, συγγνώμη, υπάρχει κόσμος άμαχος που βομβαρδίζεται από μια κυβέρνηση που θέλει να λέγεται νόμιμη. Ε, να τις προάλλες βομβαρέτησαν ένα σχολείο εκεί που ήταν μέσα από παιδιά και δέκα από αυτά ε, σκοτώθηκαν. Να, όσον αφορά την ρήτρα των δικαιωμάτων γιατί ξέρετε ότι το εμπόριο πιέζει την πολιτική. Αυτό ίσχυε από ανέκαθεν. Πάντως ε, όσον αφορά την σύντομη διαδικασία ναι Βέβαια, ε, ε, αυτό το θέλουμε ε, όλοι. Βρίσκουμε όλες τις δικαιολογίε και προφάσεις. Να σας απαντήσω σε εσά κύριε Ζαντό. Δεν πρόκειται να αντιληφθούν, να καταλάβουν οι πολίτες ότι αυτοί τους οποίους επέλεξαν δεν μπορούν να τροποποιήσουν ένα κείμενο το οποίο για ένα σωρό λόγους οδηγεί στο να υιοθετηθεί αυτή η διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι πρόκειται για μία μείζωνα εκτροπή της δημοκρατικής διαδικασίας. Δεν δικαιολογείται από τίποτε. Και αυτοί που μας ε, ψήφισαν, εμάς όλους εδώ στο κοινοβούλιο, δεν πρόκειται αυτό να το κατανοήσουν. Ο Πρόεδρος. Καλώς τώρα πολύ σύντομα η Επιτροπή, δύο συγκεκριμένα ερωτήματα διατυπώθηκαν. Παρακαλώ να δώσετε απαντήσεις. Το πρώτο ήταν αν χρειάζεται ε, παρέκκληση ΠΟΕ και δεύτερον πώς, σε, τι ύψος εκτιμώνται οι απώλειες εισοδημάτων από τους δασμούς. Απάντηση. Ευχαριστώ. Δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται παρέκκληση ΠΟΕ. Για τον ίδιο λόγο που δεν το χρειαζόμασταν και παλαιότερα φέτος, όταν υιοθετήσαμε με παρόμοια διαδικασία ε, αυτόνομα εμπορικά μέτρα, ATM. Για, και ο λόγος είναι ο εξή, το γνωρίζουν τα μέλη. Υπάρχει μια εξαίρεση των περιοχών ελευθέρων συναλλαγών από τους ε, κανόνες του ΠΟΕ και εδώ ε, θεωρούμε ότι πρόκειται περί αυτού. Όσον αφορά τώρα το, το κόστος, 78 εκατομμύρια ευρώ σε δεσμούς, στο ελληνικού δεσμούς. Αυτό μπορεί να υπολογιστεί. Αυτό που είναι πιο δύσκολο να υπολογιστεί είναι η μείωση στις, ε, στο, στο εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας, δεδομένη της πολιτικής κατάστασης στην Ουκρανία και των ε, γεγονότων, φαντάζομαι ότι το ποσό δεν θα διαφοροποιηθεί και πολύ. Αυτό που προτείνουμε αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρει. Αυτό που διαφέρει είναι ότι οι εταιρείε που από τι Ευρωπαϊκέ Ένωση που θα εξήγαν στην Ουκρανία δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αποφεληθούν από το καθεστώ το οποίο ε, διαπραγματεύτηκε η Ένωση, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά του χαμένου δασμού. Καλώ αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για το εάν θέλουμε μία απλουστευμένη διαδικασία ή όχι υπέρ μιας απλουστευμένης διαδικασίας. Κατά. Τέσσερις κατά. Αποχές. Ουδής. Απαρτία. Για την μη αποδοχή της απλουστευμένης διαδικασίας όμως υπάρχει, τέσσερις ψήφοι κατά, και ως εκ τούτου δεν προχωράει η απλουστευμένη διαδικασία, θα πρέπει να συζητήσουμε την επιταχυμένη ή την τακτική διαδικασία. Ο κύριος Κάσπαρη, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που οι φίλοι του Πούτιν και οι λοιποί δολιοφθορεί των ευρωπαϊκών ε, πραγμάτων ε, έχουν τόση παρουσία εδώ. Παρακαλώ τη γραμματεία όμως να μας δώσει μέχρι την ώρα των, ε, της συνεδρίας των συντονιστών ένα πρόγραμμα έτσι ώστε το, έως την Πέμπτη του Στρασβούργου να μπορέσουμε να θέσουμε την, έκθεση, την πρόταση αυτή σε ψηφοφορία με την τακτική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και συγχωρήστε την άγνοια του κανονισμού, αλλά όταν αρχίσαμε τη συζήτηση και ρωτήθηκε τι απαραίτητα απαιτείται, ήταν πιο λίγοι συναδελφοί εδώ. Τι εξαρτάται από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό το τι απαιτείται για να καταψήσει το κείμενο, πρόεδρος. Ναι, πρόκειται για ένα δέκατο των μελών της Επιτροπής που μπορεί να προβάλλουν τη διατήρησή τους ο κύριος Σόλτς. Θέλω απλώς στα πρακτικά να καταγραφεί η παρατήρηση του συντονιστή ε, του, Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος μίλησε για φίλους του Πούτιν. Εδώ θέλω να διαμαρτυρηθώ, γιατί δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να επηρεάζει τις θέσεις της ομάδας μου. Έχουμε, έχουμε μια αντίδραση και αντίθεση στη διαδικασία που επελέγει και αυτό θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά ο Ντάρτμορ. Θέλω απλώς να πω ότι θεωρώ πάντα πως έχω αγαστή συνεργασία, συνεργασία με τον κύριο Κασπάρη, συντονιστή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίο βλέπω ότι κρέμεται από τα χείλη μου. Η φράση ε, που άκουσα από τη Διερμηνία, φίλη των, ε, του Πούτιν και δολιοφθορείς, εάν όντως υπόθηκε, δεν έχει καμία θέση στο Κοινοβούλιο και στην ε, διαδικασία εδώ το, με, με, μου προξενεί μεγάλη λύπη αυτό. Ελπίζω ο κύριος Κάσπαρη, εν φέτο το χρόνο, να αποσύρει την παρατήρηση αυτή. Καλώς λοιπόν κλείνει εδώ η συζήτηση. Είμαστε στα διάφορα, δεν βλέπω να στα έκανε το λόγο. Προσοχέ σημείο 14 για την προσεχή συνεδρίαση 5 και 6 Νοεμβρίου που ίσως να ε, της οποίας ίσως να προηγηθεί και μια έκτακτη συνεδρίαση. Καλώς ευχαριστώ και παρακαλώ πλην συντονιστών και λοιπόν μελών να αποχωρήσετε από την αίθουσα.